Dear colleagues, we... Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ξεκινώ αμέσως με το σημείο επαριθμών 1. Έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται χωρίς αλλαγές. Σημείο 2. Οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου να σας ενημερώσω για την αποστολή της Επιτροπής ΕΝΒΗ με έγγραφα όπου έχουμε την επίσκεψη στο COP20 στη Λίμα Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τον ε, Φεβρουάριο. Στις 8 Ιουνίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου, θα έχουμε την επόμενη παρουσίαση από τον Επίτροπο Άνδριου Κάιτης για τους Γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς και θα έχουμε και μια μεικτή δημόσια κράση με την Επιτροπή ΕΝΒΙ και είτε στην, ε, στις 22 Ιουνίου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες και ως συνήθως θα μεταδοθεί και στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. για τις συστάσεις των συντονιστών 28 ε, Μαΐου και τους ε, συντονιστές έχουν ε, μοιραστεί ηλεκτρονικώς. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Και περνάμε τώρα στο σημείο 4. Ενημέρωση για τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις Μεσαίο μεγέθους μονάδες καύσης και τα νέα τρόφιμα. Για το πρώτο σημείο, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε τον πρώτο άτυπο ανεπίσημο τριμερή διάλογο με συμμετοχή του Συμβουλίου Επιτροπής και Κοινοβουλίου για σημαντικότητα για τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση. Υπάρχει σοβαρή απόσταση μεταξύ κάποιων ε, πτυχών του θέματος και θα πρέπει να υπάρξει στο δεύτερο τριμερή διάλογο περισσότερος τεχνικός συντονισμός στις, στις 2 Ιουνίου για τα νέα τρόφιμα. Όπως θα θυμάστε αποφασίσαμε την περασμένη φορά στον πρώτο γύρο τριμερούς διαλόγου αποφασίσαμε να κάνουμε πρόταση προς το Συμβούλιο για τις δύο βασικές πτυχές που ως τώρα παρέμεναν ανοιχτές. Πρώτα απ' όλα τις κατοίκους της πράξης για τον κατάλογο των νέων τροφίμων και ταυτόχρονα έχουμε και το θέμα της κλωνοποίησης. Θα πρέπει να δούμε αν θα έχουμε ένα άρθρο, μια αιτιολογική σκέψη και η πρόταση που βάλαμε σχετικά στο Συμβούλιο απορρίφθηκε. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση στη δεύτερη ανάγνωση για τα θέματα αυτά. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5. Όρια εκπομπών και έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης που προορίζονται για μη ειδικά κινητά όχι, μηχανήματα. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης από την εισηγητριά μας, την κυρία Γκαρντίνη και ευθύ αμέσως να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να θυμίσω ότι έχουμε έναν κανονισμό που υποκαθιστά τον κανονισμό 97-68 που είχε προτείνει η Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο και με τον κανονισμό αυτό θέλουμε να διαθετήσουμε τις ε, ρυπένουσες, ρηπογόνες μάλλον εκπομπές των ε, μη ειδικών κινητών ε, μηχανημάτων και προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία εναρμονισμένη αγορά στο μέγιστο δυνατό βαθμό με συγκεκριμένες προδιαγραφές παραγωγής που να αντιστοιχούν σε αυτές των πολιτείων. Εδώ κοιτάζουμε ρυθμίσεις που να ε, διδετούν τις διάφορες κατηγορίες που δεν ήταν σαφείς στον προηγούμενο κανονισμό, ιδίως για τους κινητήρες Ε, για κινητήρες που ξεπερνάνε τα 32 ΜΒ και είναι κάτω των 58 ΜΒ και για τους κινητήρες της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Ε, για τα μη κινητά μηχανήματα μας ενδιαφέρει πώς θα χρησιμοποιηθούν και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμα τις επενδύσεις. επενδύσεις. Ξεκινώ λέγοντας ότι η πρόταση της Επιτροπής συνολικά μας βρίσκει σύμφωνους είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις και μπορεί βεβαίως να βελτιωθεί όπως οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του τομέα και κάποιες κατηγορίες μηχανημάτων και κινητήρων μπορεί να καλύπτονται από τον κανονισμό. Η έκθεση που έχω υποβάλει διορθώνει 44 τοπολογίες και οι βασικότερες Ε, οι βασικότερες είναι οι εξή. Θα σταθώ σε κάποιε από αυτέ, όχι αναγκαστικά όλε, αλλά εκεί που πιο πολύ ε, μα απασχόλησε το πώς θα θετήσουμε το θέμα. Πρώτα απ' όλα για του κινητήρε αντικατάσταση. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια τέτοια ρήτρα όπως προβλεπόταν στην προηγούμενη οδηγία 97-68 για να καλύψουμε τις διαφορές σε σχέση με αυτά που ίσχυαν προηγουμένως. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ, όπως ψηφίστηκε που αναφέρεται στην ημερομηνία παραγωγής των κινητήρων, δεν μπορεί να ακολουθηθεί ως έχει, διότι για κάποιους κινητήρες μερικές φορές είναι αδύνατο να καθοριστεί η ημερομηνία παραγωγής. Όμως, ε, επί της αρχής πρέπει να πω ότι συμφωνώ όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Επίσης, η σταθερή ε, μεταβατική περίοδος 10, 15, 16 χρόνια που θα πρέπει να απολογιστεί από τη θέση σε ισχύ της κάθε φάσης εφαρμογής των μέτρων και εντός της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα υποκατάστασης ενός ε, κινητήρα ε, που θα θεωρείται αντικατάστασης, αυτό με βρίσκει θετικά διακείμενη για τις μεγαλύτερες δυνατότητες αυτή η μεταβατική περίοδος, αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο ανάλογα με κάποιους παράγοντες όπως ο κύκλος ζωής που για κάποια μηχανήματα είναι μεγαλύτερος και σε κάποιες περιπτώσεις σαφώς μεγαλύτερος. Η απόσβεση των επενδύσεων, οι, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι επίσης ένα άλλο στοιχείο που έχει να την υπόψη. Κάποιες τροπολογίες επικεντρώνονται στη μεταβατική περίοδο για να επιτρέψουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και αυτές που παράγουν και αυτές που παρά, ε, κινητήρες μόνο ή μηχανήματα και κινητήρες για να μπορούν και οι δύο κατηγορίες επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας ε, νομοθεσίας θα πρέπει να παραταθεί κάπως η μεταβατική περίοδος και να παραμείνουμε σε μια ισόρροπη προσέγγιση. Έπειτα υπάρχει ένας συγκεκριμένος τομέας αυτός των κινητών γερανών και σε ό,τι αφορά τα mobile cranes αυτά, τους κινητούς γερανούς, νομίζω απαραίτητο θα ήταν να προσθέσουμε ένα εξάμεινο στη μεταβατική περίοδο, ώστε να φτάσουμε στους 12 μήνες συνολικά για αυτή την κατηγορία μηχανημάτων και προκειμένου να καλύψουμε και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινητοί γερανοί υπόκεινται σε περιορισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις τους και ιδίως όταν μεταφέρονται οδικώς. Νομίζω ότι επιπλέον θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται για γερανούς που παράγονται και πολλούνται σε ποσότητες σχετικά ε, περιορισμένες. Ένα άλλο σημείο που με απασχόλησε είναι το όριο ως προς τις πραγματικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε σχέση με τα νέα όρια εκπομπών Βεβαίως θα υπάρξουν προβλήματα προσαρμογής και δεν θα προλάβουν όλες οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέους κινητήρε και να τους κατασκευάσουν, αλλά αν για τους μεγαλύτερους είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές, για τις μικρότερες επιχειρήσεις είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι μικρομεσαίες, οι μικρές μάλλον επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα προβλήματα ως συνήθως και επί παραδείγματι δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν όλες τις πλέον ε, σκόπιμες πληροφορίες για την δημιουργία νέων κινητήρων. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τους διατεθούν 12 επιπλέον μήνες για την μετάβαση αυτή, οι μικρές, για τις μικρές επιχειρήσεις. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων να περιληφθούν αυτές που παράγουν λιγότερα από 50 τεμάχια ετησίως, θα θεωρούσα ότι θα ήταν λογικό. Αλλά εκεί το, ανώ, το κατόριο θα μπορούσε να ε, αυξηθεί κάπως και να φτάσει στις 80 μονάδες ετησίως. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των σιδηροδρομικών. Νομίζω ότι η περίοδος ενός έτους που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να συνδυαστεί με τις υποχρεώσεις τις οποίες ήδη υπόκειται ο σιδηροδρομικός τομέας, ο τομέας των σιδηροδρόμων, άλλες νομοθετικές πράξεις όπως η οδηγία 2008-57 ε, για και ο 1302 για το τροχαίο υλικό. Ε, νομίζω εδώ ότι ο τομέας των σιδηροδρόμων θα πρέπει να εξοπλίσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κινητήρες αντικατάσταση ανάλογα με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και με συνολική αύξηση της ε, περίοδου που διατίθεται στα 15 χρόνια. Και εδώ μια πρόταση για την οποία θα ήθελα την άποψη όλων των συναδέλφων. Θα μπορούσαμε να αναβάλουμε τη θέση σε ισχύ του κανονισμού. Θα πρότεινα οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στις ε, μηχανές, τις αυτοκίνητες μηχανές να χρησιμοποιούνται και στις στις για, για την εσωτερική ναυσιπλοεία θα πρέπει να δούμε την ετήσια παραγωγή και να έχουμε μια ποιότερη προσέγγιση, ιδίω για τι πιο, για τις κατηγορίες βαρέων κινητήρων. όπως χρησιμοποιούνται για την εσωτερική ναυσιπλοεία και με ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές των ΗΠΑ. Αυτά θα μπορούσαν να συμπληρωθούν για να λάβουμε υπόψη και το ιδιαίτερο πλαίσιο εντός το κινούμαστε, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαφέρει από το αμερικανικό, ιδίω ως προς την ε, πυκνότητα της παραγωγής. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε, όπως έλεγα, τις προδιαγραφές των ΗΠΑ με τον αριθμό των ε, σωματιδίων για τους κινητήρες που ξεπερνούν τα 300 κιλοβάτ. Επίσης για μια ακόμη κατηγορία κινητήρων που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του κανονισμού για τα γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Το 167 του 13 που αφορά αυτά δεν εμπίπτουν σε αυτόν τον κανονισμό όπου μιλάμε για μειωδικά κινητά οχήματα. Αυτοί οι κινητήρες υπόκεινται σε άλλους κανόνες. Γι' αυτόν λοιπόν τον τομέα για τα τρατέ εξαρτάται από τις διαστάσεις τους για ορισμένες γεωργικές εργασίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται στους ε, οπορώνες, στα μπέλια και ούτω καθεξής. Πρέπει να προβλεφθεί ένα σύστημα after treatment και ανάλογα με το σχεδιασμό των γεωργικών ελκυστήρων δεν μπορούμε να παρέμβουμε τώρα διότι θα αλλάζαμε τις, ε, ε, δια, τις, τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δηλαδή ανάλογα με τη διαστάση τους θα μπορούσαν να περάσουν από κάποια σημεία. Είναι σημαντικό, ξέρουμε ότι τα βλάκια λόγω χάρη σε μερικέ περιπτώσει ε, αμπελιών έχουν συγκεκριμένε διαστάσει. Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε πλήρω στι διαστάσει των ΗΠΑ, όπου ίσω να μπορούσαν να προσαρμοστούν στι αλλαγέ αυτέ με διαφορετική ευκολία. Γι' αυτό στη ρήτρα αναθεώρηση νομίζω ότι καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τι ιδιαίτερε ανάγκε αυτών των μέσων. Και τέλο, τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σταθώ στην παρουσίασή μου, είναι η ρήτρα αναθεώρησης. Νομίζω χρήσιμο θα ήταν να προβλεφθεί η δυνατότητα να προβλέψουν μια πέμπτη φάση εξπόστ όπου να μπορεί το Συμβούλιο βάσει των ε, τεχνολογικών εξελίξεων και μια μελέτη κόστους ωφελίας να δει κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω μείωση των ορίων εκπομπών και να, να προταθεί σχετική ε, νομοθετική πράξη. Στην φάση 5 όμως, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και ένα ενδεχόμενο σενάριο, ώστε και όλος ο κλάδος να έχει κάτι στο οποίο να μπορεί να αναφερθεί. Ξέρουμε ότι θέλοντας να υλοποιήσουμε μια περιβαλλοντική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, δεν πρέπει παρόλα αυτά να ε, θέσουμε ένα αμφιβόλο ένα πλαίσιο βεβαιότητας εντός το οποίο ο κλάδος να προγραμματίσει και να κατευθύνει τις δράσεις του. Ευχαριστούμε και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρώτο γύρο στη συζήτηση με τους εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες Ευχαριστώ κύριε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκαρντίνη για τη μέχρι τώρα δουλειά της. Είχαμε ήδη μια πρώτη πολύ επικοδομητική συνάντηση ισχυώδης με την εισηγήτρια. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Θέλουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας και της φιλοδοξίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το πλαίσιο σίγουρα εκπομπές από το μειωδικό τομέα έρχονται περίπου στο 15% των εκπομπών αζωτούχων ε, αερίων και 5% PM είναι επομένως ρηπογόνες εκπομπές στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδίω υπάρχει για το 15% του συνόλου των εκπομπών. Το 90% λοιπόν των κατοίκων των πόλεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι εκτεθειμένη σε πολύ ψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης και γνωρίζουμε ότι πάνω από 400.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν πρόωρα επειδή εκτίθενται σε βρώμικο αέρα ε, κάθε χρόνο. Ως σκιώδης και για την οδηγία περί εθνικών ορίων Θέλω να πω ότι τέτοιου είδου νομοθετήματα είναι σημαντικά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα βέβαια όλε τι ε, πτυχέ, δηλαδή και τα, τα όρια που έχουμε σε το διάφορου όπω για την περίοδο από 2020 μέχρι 2030 για τι διαδικασίες ε, τη Κομισιόν ε, διαδικασία δηλαδή παραβάσει σε χώρες όπως μεταξύ αυτών και οι δική μου, που, χώρες που δεν πληρούν δηλαδή νομοθεσία. Σίγουρα χρειάζεται φιλόδοξη νομοθεσία αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια την ατμοσφαιρική ρήπαση. Το 2013 τα κράτη-μέλη θα ξεκολουθούν να μη συμμορφώνονται, θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους ε, και πάλι λόγω της κακής ατμοσφαιρικής ε, της ποιότητας, κακής ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα. Με συντομία, να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές της έκθεσης επί των οποίων συμφωνούμε, με κάποιες δεν συμφωνούμε. Πρώτον, μεταβατική περίοδος. Είμαστε αντίθετοι ε, σε μια περαιτέρω επιμήκυνση της μεταβατικής περίοδου για να μπορούν όλοι οι κινητήρες ε, να διατίθενται στο εμπόριο αφού τεθεί σε ισχύ το νέο πρότυπο για τις εκπομπές. Η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν 18 μήνες και ήταν για μας αρκετή αυτή η προθεσμία το πολύ πολύ ε, για μη συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να ισχύει και έχουμε ακούσει κάποια παραδείγματα που λόγω ιδιαιτερότητας ε, του μηχανήματος θα μπορούσε να έχουμε κάποια επιμήκυνση, αλλά αν καθυστερήσουμε ε, θα έχουμε πρόβλημα και με τη ρήπανση, αλλά και γιατί οι κατασκευαστές θα μπορούν να διαθέτουν στο εμπόριο πιο παλιά μηχανήματα, πιο ρηπογόνα, παρότι θα υπάρχει νέα τεχνολογία διαθέσιμη. Ε, βέβαια, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα ωφεληθούν αν επιμηκυνθεί αυτή η περίοδος και οι ΜΜΕ που δεν έχουν τους πόρους ε, για να για να αποθηκεύσουν όλα αυτά τα μηχανήματα θα πληγούν περισσότερο. Επίσης, υπό ποιε προϋποθέσεις οι εταιρείε μπορούν να αντικαταστούν, ε, έναν χαλασμένο κινητήρα. Δεν είναι πολύ αυστήρη όρη. Εγώ θα έλεγα να μειωθεί η περίοδος έγκρισης σε ό,τι αφορά του κινητήρε αντικατάσταση. Για τις περισσότερες, επίσης μια προθεσμία που προτείνει η στι περισσότερε περισσότερες ε, είναι 10 χρόνια, εγώ θα έλεγα 7. Πώς μπορούμε τώρα ε, τη διάταξη για, τις, ε, για τους κινητήρες αντικατάστασης, πώς μπορούμε αυτό να το συσχετίσουμε με κάποιες διτάξεις περί εξυγχρονισμού ε, κάποιων, ε, ε η αλλαγή κάποιων εξαρτημάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά εξαιρέσει παρεκκλήσεις είναι σημαντικό να δούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ε, να τις κρίνουμε όλες, κατά περίπτωση ανάλογα με τα και τα κατά. Αν το οικονομικό κόστος δεν είναι πολύ μεγαλύτερο από τα περιβαλλοντικά ωφέλη, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει ότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλους τους κατασκευαστέ και αν ε, για κάποιους τομείς ζητούμε λιγότερα, τότε άλλοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε όλα υπόψη. Σε ό,τι αφορά τις αοριακές τιμές εκπομπών στο παράρτημα 2, η πρόταση της Κομισιόν λίγο πολύ ευθυγραμμίζει τα πρότυπα για τα, ε, με αυτά που ισχύουν για τα βαρέα φορτηγά. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια οι και τιμές δεν είναι επαρκώς αυστηρές και θα θέλαμε να είναι πιο ε, αυστηρά αυτά τα, αυτές οι οριακές τιμές. Για, για τη φάση 3α, το 15% των συνδρομικών ε, γίνεται με διζελοκίνητα οχήματα που θα πρέπει να, είναι, να καθαρίσουμε περισσότερο. Και επίσης τα 560 κιλοβάτ και αυτή την κατηγορία ε, τα σχετικά μέτρα. Και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό υγείας και ασφάλειας, Έχουμε τροπολογία 10 συγκεκριμένα που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για κάποιους τομείς σε διάφορους ε, τόπους εργασίας. Μήπως πρέπει να επανεισαχθεί αυτή η πτυχή της υγείας και ασφάλειας στην εν λόγω νομοθεσία. Τέλος, στηρίζουμε τις τροπολογίες για την κατάσταση του συστήματος ε, έντυπης πιστοποίησης από ένα ηλεκτρονικό σύστημα, ανταλλαγή επίσης πληροφοριών, να γίνεται μέσω του συστήματος πληροφόρησης της αγοράς, είναι ήδη καθορισμένο αυτό, είναι μια λογική αλλαγή πιστεύω και με τις τροπολογίες αυτές μειώνουμε το αχρίαστο διοικητικό άρθρος και σε ό,τι αφορά την υποβολή αναφορών των αποτελεσμάτων από την Κομισιόν για τις εκπομπές. Θα πρέπει αυτό να γίνει το 2023 και όχι το 2025, αν πράγματι υπάρχουν προβλήματα αν είναι τελείως διαφορετικά πραγματικά στοιχεία. Είχαμε κάποια ε, αποτελέσματα ήδη από μελέτες για, το, για τα αυτοκίνητα, για τις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Επόμενο ομιλητή, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριο Ντάνκαν. Εμεί ε, υποστηρίζουμε την πρόταση της κυρίας Καρδίνη, εξαιρετική η δουλειά της και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να το πω αυτό. Κάνει πολύ καλά διάφορα πράγματα. Ακούσαμε τον κύριο Ντάνς ε, να λέει πόσο σημαντικό είναι να μειωθούν οι ρήποι και να συμμορφόμαστε όχι ε, μόνο προς την Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία, αλλά να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Αυτό το καλωσορίζουμε σίγουρα. Εγώ δεν θα ήμουν συντηρητικός αν δεν ε, είχα και κάποια στιγμή να σας ε, υποβάλω. Το ένα είναι τι γίνεται με τους κινητήρες αντικατάστασης και πώς θα φτάνουν στην αγορά. Το είπε και ο κύριος Ντάνς για τα οχήματα που κυκλοφορούν στο δρόμο, για το, τη διάρκεια ε, ζωής τους. Οι μικροί ε, ε, επιχειρηματίες οι αγρότες δεν μπορούν να αντικαθιστούν ολόκληρο ε, το γεωργικό τους μηχάνημα ας πούμε επειδή υπάρχει κάποια βλάβη στον κινητήρα. Ε, κάτι άλλο και χαίρομαι που και η συγγήτρια το σημείωσε και το διόρθωσε είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι αν ήταν υπερβολικά φιλόδοξοι οι στόχοι θα οθούσαν εκτός αγοράς κάποιους κατασκευαστές κινητήρων που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν, μικρούς κυρίως. Και χαίρομαι για όσα προτείνετε. Το τελευταίο που μπορεί να σας φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά αξίζει να ε, το θέσω υπόψη σας και ελπίζω να με υποστηρίξουν όλοι και οι ηγητές. Εγώ προέρχομαι από τη Σκωτία, όπως ίσως ακούτε. Περιφέρεια να την πω. Ε, χώρα, έθνος ε, που έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή και αυτό αφορά ε, ε, κάποιες λέμβους που χρησιμοποιεί η ακτοφυλακή με αξιολέμβιους κινητήρες και σώζουν ζωές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο στη δική μου χώρα. Για να γίνουν οι κινητήρες αυτοί χρειάζονται 10 χρόνια και εάν δεν ε, προσέξουμε στην νομοθεσία ενδυνεύουν να βρεθούν εκτός αγοράς. Ε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν ε, στις προδιαγραφές γιατί υπάρχει πολύ δύσκολη τεχνολογία για να ψυχρανθεί ο κινητήρας και δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Θα μπορούσα να το συζητάω για ώρες αυτό το θέμα, αλλά δεν θέλω να δοκιμάσω την υπομονή σας. Ε, θα κάνω μια τροπολογία. Αν ε, θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες είμαι στη διάθεση για να σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ από τους φιλελευθέρους, ο κύριος Βίτεμα. Στα αγγλικά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια ήταν πολύ ρεαλιστική η προσέγγιση της, την οποία εκτιμούμε και πολύ επικοδομητική άλλωστε ε, απέναντι στους υπολείπους και συγητές. Πάνω κάτω συμφωνώ απολύτως με τη γραμμή της. Και θα πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αλλά και κατά συνθήκες και κατά τομείς ε, και δραστηριότητες της οικονομίας και τι θέλουμε να κάνουμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ξανάρθει ρήτρα για ε, τους κινητήρες αντικατάστασης. Δεν μπορείς να πετάξεις ένα ολόκληρο μηχάνημα επειδή έχει χαλάσει ο κινητήρας αυτό θα έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση ε, για το περιβάλλον. Και επίσης για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει πάντα κατά περίπτωση να βλέπουμε και να προβλέπουμε ένα αρκετό χρονικό διάστημα για να προχωρήσει η καινοτομία, για την βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό επίσης να φροντίσουμε να ε, βρούμε ένα λογικό κατόφλι, μια λογική οριακή τιμή και να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τις μικρές επιχειρήσεις αλλά και τις μεσές. Και για τις κάτω χώρες έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι γίνεται με τα σκάφη της εσωτερικής δαυσιπλοείας, τα ποταμόπλια ε, και ποιε είναι οι προδιαγραφέ με τρίτες χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πολύ σημαντικό να συμμορφωθούμε προ τι προδιαγραφέ Αυτά. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία με του Σκιώδες. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Έκο, κύριο Σεκχάουτ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Καρδίνη για την ε, δουλειά της σε αυτό το θέμα. Αναφέρθηκε μια-δυο φορές, είναι ζωτική σημασία. Και παρόλο που ακούγεται πολύ τεχνικό, πρέπει να εξηγήσω τι συμβαίνει με τον κανονισμό αυτό και με τις τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει. Γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω κάτι στον συνάδελφο από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστές, Διότι αυτή τη στιγμή έχετε αναλάβει την έκθεση για την οδηγία ΝΕΚ που ορίζει τα όρια. Και όποτε έχουμε διαπραγματεύσει με τον συγγήτρια από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, μα λέει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καλή νομοθεσία για το επίπεδο των ε, πηγών. Διότι αν προβλέψουμε ένα ανώφλι και αν έχουμε κοινό επίπεδο για όλε τι πηγέ, θα είναι πολύ δύσκολο να σεβαστούμε αυτό το ανώφλι, το ανώτατο όριο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πηγαίνει και θα λέει στι χώρε ότι δεν συμμορφώνονται. Και υπό αυτήν την έννοια βλέπουμε το συσχετισμό οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ διαρκώ επιμένουν στην πολιτική για τι πηγέ. Εδώ την έχουμε στα χέρια μα την ευκαιρία. Τι κάνουν οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ, καθυστερούν την υλοποίηση και ζητούν όλο και περισσότερε εξαιρέσει. Δεν είναι πάρα πολύ συνεπή η στάση σα. Εφόσον πάντοτε επιμένετε για την καλύτερη νομοθεσία, τουλάχιστον αρχίστε να δείτε, γυρίστε και κοιτάξτε τι γίνεται στην δική σα εσωτερική νομοθεσία και κατά πόσο εκεί είστε συνεπεί πριν οδεύσουμε στην κατεύθυνση της ε, αύξησης των ε, εξαιρέσεων και της ε, βραδύτερης υλοποίησης, ας φροντίσουμε να μην είμαστε τουλάχιστον ασυνεπείς όταν ορίζουμε τα ανώτατα όρια για τα διάφορα ειδηρήπων, τα ζωτούχα και ούτω καθεξής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Δεν θα σας εκπλήξει, κυρία Γκαρντίνη, που θα έχω απαιτητικά σχόλια για την έκθεσή σας, παρόλο που εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά σας, όμως έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί η φάση της υλοποίησης να παραταθεί και να πάει από 18-24 μήνες και γιατί να προβλεφθούν προφανείς εξαιρέσεις με τις τροπολογίες 16 και 17. Επίσης, μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των εξαιρέσεων αυτών. Θα ήθελα λίγο περισσότερες εξηγήσει. Ε, δεν το προτείνατε εσείς έτσι και πριν ε, συζητήσουμε τις εξαιρέσεις αυτές που δεν τις βλέπουμε θετικά, θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αντίκτυπο εκτιμά ότι θα έχουν αυτές οι εξαιρέσεις ε, και τι προσπαθεί να επιτύχει εδώ. Ιδάλλως, πάλι φτιάχνουμε ένα τυρί με τρύπε, δηλαδή νομοθεσία με παραθυράκια, που ε, κάποιοι από τη δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου θα αρχίσουν να το επικρίνουν και να λένε ότι είναι δύσκολο να το υλοποιήσει κανεί. Το ίδιο και για το τυρί. Μπορεί κανεί να αποφύγει τι τρύπε αν φροντίσει από την αρχή τη Παρασκευή του να μην υπάρχουν. Πάντω, ε, να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε την νομοθεσία. Ναι, αλλά πάρα πολύ προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε με τι ΗΠΑ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το TTIP, φαντάζομαι, έτσι, και τι διαπραγματεύσει του. Ερώτηση σα θέτω. Είναι πραγματικά ε, εκπληκτικό να βλέπουμε ότι σε κάθε νομοθεσία που προβλέπουμε πλέον ε, φροντίζουμε να ευθυγραμμιζόμαστε σε όλα με τι ΗΠΑ. Ε, και λένε πολλοί ότι δεν θα επηρεαστούν οι νόμοι που εμεί εγκρίνουμε τώρα από τι διαπραγματεύσει TTIP και τη συμφωνία. Τότε γιατί να μην ευθυγραμμιστούμε με την Ελβετία, μια χώρα που είναι σε ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση για τι εκπομπέ, την, ε, τα όρια για τι εκπομπέ. Γιατί δεν κοιτάζουμε αυτή τη χώρα που είναι μπροστά και κοιτάζουμε τι. ΗΠΑ. Και θα μπορούσε η υλοποίηση να προχωρήσει και πολύ πιο γρήγορα ε, από ό,τι ορισμένοι εδώ δηλώνουν. Νομίζω λοιπόν καλύτερα να κοιτάμε τους πρώτους παγκοσμίω και όχι του τελευταίου. Ε, και ε, αν μπορείτε, επιβεβαιώστε μου ότι καμία σχέση δεν υπάρχει με τι του τη συμφωνία TTIP. Κάτι που έχει εξηγηθεί ε, ξανά και ξανά και ξανά και αρχίζω να μην σας... Πολύ πιστεύω κιόλα πρέπει να ομολογήσω. Και για να ολοκληρώσω, ε, ανυπομονώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, να είστε βέβαιοι ότι θα κοιτάξω να είμαστε πολύ συνεπέστεροι με αυτά που επιδιώκουμε στην οδηγία αυτά που επιδιώκουμε στην οδηγία ΝΕΚ και επιπλέον ελπίζω να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια, αλλά είστε βέβαιοι ότι αν ε, συμφωνήσουμε για τι περαιτέρω εξαιρέσει και παρατάσει τη περίοδου, υλοποίηση, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε επιχειρήματα που να σταθούν και για την ώρα δεν έχω ακούσει τέτοια. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η κυρία Εμπι Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Παρά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λείπουν κάποιες ε, παράμετροι όπως για τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα και οι χρόνοι υλοποίησης δεν φαίνονται αρκετοί για την προσαρμογή στις νέες προδιαγραφές. Ορισμένε προτάσει εξαιρέσεων, όπω προτείνονται από την εισηγήτρια, δεν μα ε, πείθουν πλήρω, όπω και από ένα επαναπροσδιορισμό των ε, νέων κατηγοριών και των ε, όσων προβλέπονται στο παράδειγμα 2 και 3 υπάρχουν και ορισμένες τροπολογίες με στόχο τον εξορθολογισμό διοικητικού κόστους ε, ε, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κατομελών και εκεί μας βρίσκουν σύμφωνος. Το ίδιο και η ιδέα να μπορούμε να υποκαταστήσουμε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με ε, τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται με ηλεκτρονικούς κώδικες στην σχετική βάση δεδομένων. Πάντως θα είναι χαρά μας να ε, συνεργαστούμε για την ε, τελική μορφή της έκθεσης, παρόλο που εδώ συμμερίζουμε τις ανασυχίες του συναδέλφου Eckhout. Δηλαδή η διαρκής παρουσία των ε, Ηνωμένων Πολιτειών ε, αναφέρεται συχνά στην αναθεώρηση της οδηγίας αυτής και στο γιατί τους επιλέγουμε ως πρότυπο. Και εγώ συμμερίζομαι αυτές τις αμφιβολίες. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκροστέ τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μου, την κυρία Γκαρντίνη, να τη εκφράσω την υποστήριξή μου για την έκθεσή της εν Θα ήθελα ωστόσο να επιμείνω σε ορισμένα σημεία. Μεταξύ αυτών σε κάποια που αφορούν το συνδρομικό τομέα, ίσως γιατί στη Γαλλία αυτή τη στιγμή πραγματικά συζητάμε πολύ τα περί του συνδρόμου, πώς εξελίσσεται η κατάσταση στον τομέα αυτό και αυτό και στρέφουμε πιο πολύ εκεί. Ε, βέβαια, το 80% των σιδηροδρομικών μεταφορών γίνεται με ηλεκτροδότηση, ηλεκτροδοτούμενες γραμμές. Υπάρχει όμως και ένα 20%. Εκεί ε, παραμένουν κάποιες ε, σιδηροδρομικές μηχανές που είτε λόγω έλλειψης υποδομών, είτε γιατί δεν αντικαταστάθηκαν, έχουν μηχανές diesel, κινητήρες diesel. Το diesel είναι σαφές ότι πρέπει να αντικαταστάθει το συντομότερο δυνατό για λόγους ποιότητας βέβαια του ατμοσφαιρικού αέρα και για λόγους υγείας, όμως υπενθυμίζω ότι από τη στιγμή που θέλουμε να εμφαρίνουμε τις δρομικές εμπορευματικές μεταφορές σε μια χώρα όπως στη Γαλλία για παράδειγμα, ήδη πρέπει να σας πω μάλλον ότι ακόμα υπάρχουν δυσκολίες ε, σε σύγκριση με τη μεταφορά εμπορευμάτων ε, οδικά, θέλω να πω προσοχή συνάδελφοι. Συμφωνούμε, ναι, πρέπει να υπάρξει πρόοδος, αλλά χωρίς να μπούμε σε μειονεκτική θέση. Με ανησυχούν τα άρθρα 3.31, 31, 3, 4 για αντικατάσταση των δηλοκινητήρων μέσα σε πολύ σύντομες για μένα χρονικά προθεσμίες. Αυτές οι προθεσμίες είτε για τους βιομηχάνους είτε για τις συνδρομικές εταιρείες δημιουργούν πρόβλημα, διότι οι συνδρομικές εταιρείες έκαναν επενδύσεις μακροπρόθεσμες, πρέπει να προσαρμοστούν, αλλά πρέπει να έχουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Κατά την άποψή μου λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι για την αντικατάσταση των διζελοκινητήρων αυτών και γι' αυτό στηρίζω τις προτάσεις της Ελιζαμπέτα Γκαντίνη με τις τροπολογίες 16 και 17. Τώρα, το άρθρο 57 της πρότασης της Κομισιόν προβλέπει μεταβατικές περιόδους, μίλησαν κάποιοι συνάδελφοι, διάρκεια 12-18 μηνών για την αντικατάσταση μηχανημάτων και κινητήρων που κυκλοφόρησε τον εμπόριο αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικές αυτές οι προθεσμίες. Αν βάλουμε το χρόνο που χρειάζεται μόνο για την ε, σύναψη των συμβάσεων, για την προκήρυξη διαγωνισμών, που ξέρουμε πόσο αυστηρά είναι τα όρια, δεν γίνεται δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια προθεσμία. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε περιόδους ε, τη τάξη των 18-24 μηνών. Αυτέ είναι ρεαλιστικές προθεσμίε. Συμφωνώ και χαίρομαι μάλιστα που η συγκήτρια κάνει ρεαλιστικέ προτάσει. Αυτά συγκεκριμένα για την έκθεση κυρία Γκαρντίνη θα καταθέσω τροπολογίε, αλλά γενικά εξαιρετική δουλειά τη βρίσκω. Σας ευχαριστούμε, η κυρία Πύρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκαρδίνη. Όλα πράγματα που μου υπέβαλαν και από την Ολλανδία για γεωργικούς ελκυστήρες και άλλα τα έχετε συμπεριλάβει πάρα πολύ καλά. Ένα σημαντικό στοιχείο που το είπε και ο συνάδελφος Γιάν Χαϊτεμα έχει να κάνει με την εσωτερική ναυσιπλοεία. Ε, ε δείτε και σε σχέση με το σιδηρόδρομο είναι πολύ σημαντικά αυτά. Τα έχετε ε, θεωρήσει κι εσείς. Μιλάτε για ευθυγράμμιση με τα αμερικανικά πρότυπα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν θα κάνω τροπολογίες, αλλά δεν νομίζω ότι εντάσσεται απόλυτα σε αυτό το κανονισμό, αλλιώς να κάνω τροπολογία. Μας είπαν κάποιοι κατασκευαστές κινητήρων ότι θα πρέπει να, αν πρέπει να ευθυγραμμιστούμε όλοι στα αμερικανικά πρότυπα, δεν θα μπορέσει ο δικός μας κλάδος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό στην Ολλανδία, να προσαρμοστεί. Ευχαριστώ. Thank Θα δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Εσκομπάρ Γκερέρο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει η Κομισιόν για την πρόταση αυτή της κυρίας Γκαρντίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το οικοδομητικό έργο που έχει επιτελέσει και για τα αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε. Με βάση τη δική μας αντίληψη η πρόταση ως έχει ε, και όπως συζητείται και στο Κοινοβούλιο αλλά και στα κράτη-μέλη και από τις συζητήσεις φαίνεται ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων οπότε πιστεύω ότι τελικά θα σημειώσουμε πρόοδο και θα έχουμε ένα ρυθμιστικό κείμενο που θα μας επιτρέπει να τηρήσουμε φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους αφενός, αλλά και να διατηρήσουμε και τους στόχους αστικής αγοράς αφετέρ. Τέσσερα σχόλια, τέσσερις ομάδες σχολείων. Καταρχάς, συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγής σε πληροφοριών πιο σύγχρονο. Αυτό το θεωρούμε καλό δείγμα, καλό ιονό. Ε, δεύτερον, που θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ανοιχτοί και συνεργάσιμοι όπως ήδη κάναμε και στις συζητήσεις ε, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Καταρχάς αυτό αφορά διατάξεις όπου οι συγκεκριμένα στοιχεία διατάξεων αφορούν την εσωτερική ναυσιπλοεία, τους όρους για τις κινητήρες αντικατάστασης, τις κινητήρες που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρόμους, που είπε και η κυρία Γκροστέτ, και της ρήτρας την αρχή της δεύτερης αναθεώρησης. Έχουμε όμως και κάποιες δυσκολίες, όπως αφο... για παράδειγμα ε, σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις ή την επιμήκυση μεταβατικών περιόδων. Με βάση την ανάλυση μας, αυτό θα ήταν παραγωγικό σε σχέση με τη διαχείριση των αποθεμάτων για τους παραγωγούς αλλά και για τους ε, χρήστες. Τρίτο στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει με κάποια άλλα θέματα που αναφέρθηκαν. Κάποιοι βουλευτέ ρωτούν για το retrofitting γιατί δεν έχουμε κάποια διάταξη. Πράγματι έχουν μια δυσκολία γιατί μιλάμε αποκλειστικά για τα προϊόντα τα οποία διτίθενται στο εμπόριο. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να δούμε και πάλι κάτι που είχε προτείνει η Επιτροπή για τις εκπομπές για τα φορτηγά. Οπότε είχαμε εκεί κάνει κάποιες ε, σκέψεις και ότι, σε ό,τι αφορά αυτές τις μετατροπές, το retrofitting, είχε κάνει κύριος Γκρότη κάποιες προτάσεις τότε, όπως για παράδειγμα κοινά κριτήρια. Μπορούμε να έχουμε κοινά κριτήρια για να βάλουμε τις διατάξεις περί μετατροπής στην εθνική νομοθεσία. Θεωρήθηκε φρικτό να μπουν αυτές οι διατάξεις σε ένα κείμενο που νομίζω ότι είναι και σχετικά παρόμοιο με τις εκπομπές, με το κείμενο που αφορά τις εκπομπές των μηχανημάτων. Τώρα, η σχέση αυτών των διατάξεων με τα αμερικανικά πρότυπα, ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι το μοντέλο που ακολουθήσαμε είναι το μοντέλο των αμερικανικών κανόνων και προτύπων από τα οποία κάποια θεωρήσαμε χρήσιμα, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο παραδείγματος για τα σωματίδια. Εκεί είπαμε ευθύ αμέσω και νομίζω ότι συμφωνείτε, ότι δεν είναι ικανοποιητική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα λεπτά αυτά σωματίδια στην Αμερικανική νομοθεσία. Πρόταση τη Κομισιόν λοιπόν είναι να δούμε τι λειτουργεί στην πράξη. Κάποια πρότυπα θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα, για κάποια δεν έχουμε την διάποψη. Δεύτερον, κάναμε μελέτη αντικτύπου. Πριν από οποιαδήποτε συζήτηση επί Ουσιαστικά αναλύσαμε ποια είναι τα πλέον κατάλληλα πρότυπα. Και το τρίτο, σας ενημερώνω ότι εξ όσο γνωρίζω, τουλάχιστον εγώ, δεν γίνεται κάποια συζήτηση σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο για αυτά τα πρότυπα στο TTIP. Άρα συζητάμε τα υπέρ και τα κατά και την ανάγκη να έχουμε επίπεδα εκπομπών που αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες αλλά και στις ανάγκες προστασίας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γκαρντίνη, για την ε, καταληκτική της παρέμβαση. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο τους σκιώδεις συζητητέ, με τους οποίους ήδη ξεκινήσαμε μία συνομιλία πολύ ε, επικοδομητική, πραγματιστική και ε, έντονη συνεργασία. Όλοι έχουμε κοινό στόχο, όπω το θύμισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να προβλέψουμε νομοθεσία που θα προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία και ταυτόχρονα και την κοινή αγορά. Είμαστε σε μια συγκυρία που μα το απαιτεί. Μα το απαιτεί κατά απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε το σημείο αυτό μέγιστης προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας έχοντας ως προτεραιότητα ακριβώς την ε, υγεία και το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Άρα χωρίς να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κλάδο πολύ ποικίλο και με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και που ήδη έχει συμβάλει τα μάλα στην συνολική ρήπανση όπου ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι επιμέρους κλάδοι πρέπει να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους και συνολικά να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ε, γιατί έχουμε κάποιες περιπτώσεις ρήπων που φτάνουν το 90-95%. Μιλούμε λοιπόν για κάποια αριθμητικά στοιχεία περιθωριακά μεν, αλλά ε, ουσιαστική σημασία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εκείνο το σημείο που θα προσφέρει την ανάλογη ισορροπία ώστε να μην έχει και αντίστροφε συνέπειε στο περιβάλλον για του σιδηροδρόμου. Ε, το 90% των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ηλεκτροκίνητε. Όμω το 20% είναι διζελομηχανέ αυτό ε, ε, αφορά κυρίως επαρχιακές γραμμές ορεινών περιοχών όπου η ηλεκτροκίνηση δεν είναι τόσο απλό να εφαρμοστεί. Το να το επιβάλλουμε θα πει ότι θα καταργήσουμε τελείως κάποιες σιδηροδρομικές γραμμές και θα πρέπει να την καταστήσουμε με τις οδικές. Κάτι που θα είναι ακόμη πιο ρηπογόνο. Ε, αυτό έχω κατά νου όταν λέω να οθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εκεί που γνωρίζουμε ότι θα έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα υπενθυμίστηκε και νομίζω ότι όλα τα σημεία που ε, αναφέρθηκαν πρέπει να τα μελετήσουμε ένα προς ένα. Το ίδιο προς τον συνάδελφο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που λέει ότι θα προτιμούσε τα χρονικά διαστήματα να είναι 7 ε, τα χρόνια αντί για 10. Θα το μελετήσουμε συγκεκριμένα, διότι αν η επταετία είναι καταλληλότερη από τη δεκαετία, καλύτερα, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, όμως ας ε, πάρουμε, ας, δούμε μάλλον αν μπορούμε να μελετήσουμε από κοινό όλες τις προτάσεις που έγιναν σήμερα για να βρούμε μια πραγματιστική πρόταση και να αντιποκριθούμε και στις ανάγκες της πραγματικότητας. Αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να εντοπίσουμε την σωστότερη προσέγγιση. Να βρούμε τον ορθότερο ορισμό στον κανονισμό αυτό, εντοπίζοντας τα σωστά όρια και τα σωστά χρονικά διαστήματα. Να θυμίσω ότι εδώ ομιλούμε για τομείς και κλάδους ε, ιδιαίτερους. Μιλούμε για μηχανήματα που έχουν κύκλο ζωής πολύ μεγάλο πολλές φορές, αλλά έχουμε έναν κλάδο, ένα τομέα πολύ ποικίλο, με μεγάλες διαφορές του κύκλου ζωής. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να έχουμε το χρόνο, σε αυτή την εβδομάδα, αυτέ τι ημέρε να μελετήσουμε αναπερίπτωση το τι συμβαίνει για να βρούμε τη σωστή, ε, το σωστό προγραμματισμό. Εδώ μιλάμε και για παραγωγού. Δεν ξέρω εάν σωστά ερμήνευσε αυτό που ο συνάδελφο των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών που λέει ότι λείπει η διαδικασία διευθέτηση του κύκλου ζωή των μηχανημάτων, των οχημάτων μάλλον. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα σημαντικό θέμα που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη τη στιγμή που ε, θα προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε το τι κάνουν οι παραγωγοί, αλλά μην ξεχάσουμε ότι με αυστηρά όρια μπορεί, όπως ήδη συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να παρατείνουμε το σύνολο, την, το κύκλο ζωής ενός ρηπογόνου στόλου οχημάτων και τελικά να έχουμε το αντίστροφο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν θα απαντήσω σε όλους έναν προς έναν. Σας ευχαριστώ. Σημείωσα όλες σας τις παρατηρήσεις, όλα τα σχόλια και νομίζω ότι ε, είναι ουσιαστική σημασία. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας, την κοινή δουλειά που κάνουμε όλοι μας και μας έχουμε ακριβώς καλή τύχη. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Ε, προθεσμία για την υποβολή 4 Ιουνίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΝΒΗ 15 Ιουλίου και θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα δίλεπτο και μετά θα ψηφίσουμε. Dear colleagues, we can... Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πρώτο σημείο, σημείο 6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106. Αφαίρεση ορισμένων αρωματικών ουσιών από τον κατάλογο της Ένωσης. Ε, μία και μόνο ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. περιμένουμε. Ωραία. να απαντήσω. Πέρα τη ψηφοφορίας. Ok, il voto è chiuso. No. Ok, il voto è chiuso. Peras. Απορρίπτεται. Πάμε στο σημείο 7. αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς. Ονομαστική ψηφοφορία, ηλεκτρονική δηλαδή, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Αγκρίνεται. Ascoltiamo adesso il... Ψηφίζουμε την έκθεση της συναδέλφου Χέραντ Καρσία για τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες. Ξεκινούμε με τη συμβαστική 1. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 τη συναδέλφου Ριβαζή. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Εβδομήντα τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 του συναδέλφου Ρεβαζή. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Δεν ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνατε. 18 και 81. Πανομοιότυπες. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 82. Πρώτο τμήμα. Όπως προστέθηκε στη συμβαστική 3, συγκεκριμένα τους όρους ιδιαιτέρες του πλέον ε, ευάλωτου του τμήματος της κοινωνίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. 90. 90. Επέρ. Κατά. Αποχέ αγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92. Με συγχωρείτε, 93. 92. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους σοσιαλιστές. Δεν σηκώνουν τα χέρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Εψήφισαν πέρας. Εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. ξανά άπαντες πέρας. Αγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έξι άπαντες. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται έλεγχος. Εψήφισαν πέρα πέρας. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 και 32 πανομοιότυπες υπέρ κατά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 κατά απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. ξανά άπαντες. Πέρασε. Εμενταμέντο. Η τροπολογία υπάρχουν 44. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθμών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 50 Υπέρ. Κατά. Αποχές απορίψετε. Η 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Η τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Η 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. ψηφίπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Ή 56. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη. Ή 57. Υπέρ. Κατά έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Ε, εγκρίθηκε. Η τροπολογία παριθμό 58. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία ειναι 9. Πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά έλεγχος. Avete Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 64 ψήφιπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 65 με μια προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ. Διαφωνεί κανείς. Αλλιώς δεν θα το ψηφίσουμε. Υπέρ δεν διαφωνεί κανείς. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την τελική πρόταση όπως τροποποιήθηκε αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ε, ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Dobbiamo fare il voto sulla ε, Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ε, παρακαλώ τους συναδέλφους που θέλουν να αποχωρήσουν να το πράξουν. Ε, ε, Πάμε στο επόμενο θέμα. Αποτελεσματική χρήση των πόρων μετάβαση σε μια κεκλική οικονομία. Είναι η εξέταση των τροπολογιών. Στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης θα δώσω αμέσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Πιετικάινεν για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες και να τις σχολιάσει. Παρακαλώ κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν αρκετά πολλές, ε, γύρω στις 400 και κάτι. Όταν όμως μετά τις ε, εξετάσαμε μία προς μία, τις και κάποιες από αυτές ε, δεν χρειάστηκε να τεθούν σε ψηφορία τελικά. Μιλάμε λοιπόν ε, για αυτούς τους μευτικούς ε, πόρους. Ε, κάποιοι θέλετε να είναι πιο απλοί ορισμοί, κάποιοι θέλετε να είναι πιο αυστηροί κτλ. Ένα άλλο σημείο είναι, και αυτό το βλέπετε σε διάφορα σημεία της έκθεσης, κατά πόσο πρέπει να γίνεται ε, εθελοντικά, να γίνονται εθελοντικά κάποιες ενέργειες ή νομοθετικές πράξεις να θετούνται. Εγώ είμαι σάβος ότι το εθελοντικό δεν αποδίδει, είναι σαν να πληρώνει κανείς εθελοντικά φόρους. Και δεν είναι και ισότιμο πεδίο ε, ανταγωνισμού για όλους τους φορείς. Υπήρξε επίσης κάποιες καλές τροπολογίες ό,τι αφορά την ποιότητα του ιδιωτικού δυναμικού και ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Πολλοί λόγος έγινε για τους δείκτες, αν πρέπει να είναι δεσμευτικοί ή όχι, αν πρέπει να είμαστε λεπτομερικοί και να περιλάβουμε και επιμέρους δείκτες. Εγώ νομίζω ότι καλό είναι να είναι πιο γενικοί οι δείκτες και όχι να αναφέρουμε συγκεκριμένα ε, το νέο και κάποιους άλλους δείκτες ξεχωριστά. Οι στόχοι επίσης έγιναν αντικείμενο συζήτηση αν θα είναι δεσμευτική ή όχι. Και όπως και στην περίπτωση λογιστικής ε, πιστεύω ότι από τη στιγμή που το κάνουμε πρέπει να είναι υποχρεωτικό για να υπάρχουν ε, κοινά κριτήρια, αλλιώς δεν έχει νόημα να προωθήσουμε μια τέτοια νομοθεσία εάν επιτρέπουμε εθελοντικά να γίνονται ορισμένα πράγματα. Ε, Επίσης έχουμε κάποιες σημαντικές πρώτες αναφέρονται κάποιες τέτοιες πρώτες ύλε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα έχουμε βιώσιμα κτίρια ε, και βιώσιμα τρόφιμα. Λόγω του περισμένου ε, χώρου, νομίζω ότι καλό είναι να είμαστε γενικόλογοι και να μην ε, αναλύσουμε τους διαφόρους τομείς. Όχι ότι έχω και κάτι βέβαια κατά, επί της αρχής. Σε ό,τι τώρα επικίνδυνες ουσίες ή το στόχο για την ε, εξάλληψη διάθεση τοξικών χημικών ουσιών. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Και βέβαια πολλές τροπολογίες όπως φαντάζεστε για τα μηδενικά απόβλητα. Αυτό το στόχο και την σχετική οδηγία. Και η ανάγκη για την οδηγία περικολικού σχεδιασμού. Δεν ε, θέλω να καταλήξω κάποια λάθος συμπεράσματα, αλλά όπως καταλαβαίνω Πολλές τροπολογίες μπορούν ε, να συμπεριληφθούν χωρίς πρόβλημα, αλλά έχουμε και κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει διάσταση απόψεων. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε με κάποιες συμβαστικές προτάσεις να βρούμε τη μέση ε, οδό, τη χρυσή τομή. Θα το συζητήσω με τους σκιώδεις συγητές και ελπίζω να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις. Αν έχετε ερωτήσεις ε, ή υποδείξεις, ε, κριτικές, ε, ευχαρίστως να αντιδράσω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for your... Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Αρχίζουμε λοιπόν. Πρώτα με τους σκιώδεις συγητές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζόφολη που θα μιλήσει εξ με του κύριου Παολούτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Παολούτσι. Εκείνος κάποια στιγμή θα σας παρουσιάσει τις τροπολογίε και τις συμβαστικέ, αλλά ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία γενικού χαρακτήρα και μετά σε μερικέ παρατηρήσει για το τμήμα που αφορά τα απόβλητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιτρόπου Σεύκοβιτ επιβεβαίωσε ότι εντό του 2015 θα πρέπει να υποκληθεί μια πρόταση για την αναθεώρηση τη οδηγία για, την, ε, συμβατή, για τον οικολογικά συμβατό σχεδιασμό και για, τα, για τον εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια. Ζητούμε αναθεώρηση τη οδηγία αυτή να συμπεριλάβει όχι μόνο τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, αλλά και τα κατασκευαστικά υλικά, τον εξοπλισμό και την επένδυση για να δώσω και την ένδυση, για να αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. Ω προ την αναθεώρηση που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να ορίσουμε και ελάχιστε τιμέ για τα υλικά που ανακυκλώνονται και θα χρησιμοποιούνται στα νέα προϊόντα. Μία άλλη παρατήρηση αφορά όλο ιδιαίτερω τα θαλάσσια απόβλητα. Βάσει των δεσμεύσεων που αναλάβαμε στο Ρίο 20, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει έναν ε, δεσμευτικό στόχο και για αυτό το είδο τα απόβλητα. Μία μείωση το 50% εντό του 2025 λόγω χάρη με απαγορεύση κάθε απόρριψη πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα και υλοποιώντα τη Διεθνή Σύμβαση Μάρπολ για την πρόληψη τη ρήπανση που προκαλούν τα σκάφη. Μια άλλη γενική παρατήρηση. Ε, συμμεριζόμαστε την ε, πλήρη ε, σωρευτική χρήση των ε, πόρων όπως την ξυλία αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην βιομηχανική χρήση της βιομάζας στην ιεράρχηση της αποκομιδής αποβλήτων ιδίως για το μείζο μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Τέλος, συμφωνούμε με την εισαγωγή δεσμευτικών δικτών για την κατανάλωση όχι γενικώ και ορίστος των πόρων, αλλά πολύ συγκεκριμένα για την, ε, για την κατανάλωση νερού, για την ε, αποκομιδή των απορριμμάτων στο έδαφος και για να καλύψουμε και τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, όχι μόνο τις περιβαλλοντικές, στις οποίες πρέπει να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξωευρωπαϊκές της διαπραγματεύσεις με τις εκτός ένωσης χώρες και στις διεθνείς συμβάσεις, ώστε να ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές για όλους. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούνται δείκτες για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Σε ό,τι αφορά όλος ιδιαίτερο τις πολιτικές των αποβλήτων, Έχουμε υποβάλει διαφορετικές προτάσεις που θα τις ανακεφαλαιώσω. Ζητούμε η απαγόρευση στην ε, θέση σε χωματερές ε, σε χείτα των βιοδιασπόμενων ε, αποβλήτων να προβλεφθεί στο 2020 και ως τότε θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, καθορί, να επιβάλλει την διαλογή των βιοδιασπόμενων απορριμμάτων ώστε να διαχωρίζονται αυτά που προέρχονται από την κατασκευή ή από την διάλυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα είναι εντό του έτου να υποβάλει νομοθετική πρόταση ώστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, ορίσουμε στόχο 70% μέχρι το 2030 για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών αποβλήτων. Ε, μεταξύ των στόχων θα πρέπει να προβλέψουμε και έναν ορισμό με μια μέθοδο κοινού υπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια και επιστρέφουμε στις ε, χωματερές, κάποια κατάλοιπα δεν μπορούν να τοποθετούνται, να, να αποτίθενται στις ε, χωματερές, οπότε μέχρι το 2030 ζητούμε η απαγόρευση για την διασφάλιση αυτών των μη των ε, απορριμμάτων που δεν είναι κατάλληπα, να μην ξεπερνούν το 5% του, της συνολικής παραγωγής αποβλήτων και μερικές παρατηρήσεις για την ε, ενεργική αποδοτικότητα στα κτίρια. Ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει ένα πλαίσιο στόχων με ένα πίνακα που θα χρησιμοποιείται στο Ρώσιμπο, με κάποιου στόχου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τα επίπεδα που θεωρούνται βιώσιμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κάτι μέλη να προβλέψουν περαιτέρω δείκτες, ε, μεθόδου και παραμέτρους για την ε, αστική χωροταξία. Και εδώ χρειάζεται μια προσέγγιση που να είναι ταυτόχρονα ε, και περιβαλλοντικά βιώσιμη αλλά και οικονομικά και κοινωνικά. Και σε ό,τι αφορά τους ε, πόρους στην ε, κατασκευή κτηρίων θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πόρους και να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος με απαγόρευση της θέσης ε, των ε, υλικών που έρχονται από κατασκευή και διάλυση έως το 2030 και σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθεί μια στρατηγική ε, συντονισμένη και μακροπρόθεσμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανακαίνιση των ε, υπαρχόντων κτηρίων. Έτσι θα έχουν ρόλο ενισχυμένο ρόλο να διαρματίσουν και τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να προβλέψουν πρωτοβουλίε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διοικητικό. Με αποτελεσματική ανακαίνιση του ε, της κτηριακής μας κληρονομιάς. Επίσης την ε, απουσία δημοσίευσης ε, της, του καταλόγου για την βιώσιμη κατανάλωση, την επισητιστική, Καλό θα ήταν η πρόταση αυτή να δημοσιευτεί, να υποβληθεί εντός της χρονιάς ώστε να έχουμε περιορισμό της κατασπατάλησης ε, τροφίμων στο το 2030 κατά 30%. Ε, έχουμε επίγνωση βέβαια ότι αυτή η στρατηγική η στρατηγική για την κυκλική οικονομία με όλες τις πτυχές θα πετύχει μόνο αν υπάρξει εκπαιδευτική προσπάθεια με συμμετοχή όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ε, των κοινοτήτων, δήμων, περιφερειών και επαρχιών αλλά και τη ενώσης των πολιτών και επίσης θεμελιώδης σημασία είναι να επενδύσουμε στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση για να έχουμε τις απαραίτητες ε, ικανότητες που χρειάζονται από αρχιτέκτονες, εργολάβους, ε, χωροτάκτες και να ε, δώσουμε δυναμικό χαρακτήρα στην υλοποίηση της σχετικής πρότασης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ντεμισμέκερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. πάρα πολλές τροπολογίες. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον ε, του θέματος. Έχω κάνει διασκέψεις, σκέψεις, ε, έχω διέγγραφα θέσεων, έχω κάνει προγεύματα εργασίας ε, για αυτά τα θέματα. Ό,τι έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία είναι πάρα πολύ ζωντανό και εδώ στο Κοινοβούλιο και εκτός του Κοινοβουλίου. Είναι καυτό θέμα και είναι ε, πολύ θετικό που είναι στρατηγική ε, αυτή η ε, πρωτοβουλία μας και θέλουμε να την ολοκληρώσουμε πριν τις ενές διακοπές. Είναι πολλές οι τροπολογίες, είναι πολλά τα στοιχεία που έχουμε επιτάπητος και ε, θα εξαρτηθεί από την εστίαση. Δεν θα είναι εύκολο καθόλου. Θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες και να ξεκαθαρίσουμε ότι η φιλοδοξία μπορεί να ενωθεί με το ρεαλισμό στην πρότασή μας για να στείλουμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσβλέπω εδώ και στις συμβαστικές προτάσεις της εισηγήτριάς μας. Σε ό,τι αφορά την προσωπική μου θέση, ήθελα να σας ε, πότε τα εξή πέντε επιγραμματικά. Πρώτον, η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι για μένα απαραίτητη για να λειτουργήσει η ίδια μας η οικονομία με τρόπο βιώσιμο και αηφόρο. Η Ευρώπη εξαρτάτε εξαρτάται πάρα πολύ από ε, πρώτες ύλες που ε, εισάγουμε και οι δικές μας μειώνονται πάρα πολύ. Κυκλική οικονομία λοιπόν όπου θα μπορούμε να ανακυκλώνουμε υλικά και προϊόντα, να τα επισκευάζουμε, να τα επαναχρησιμοποιούμε. Ε, είναι κατεξοχήν φιλική προς το περιβάλλον αλλά μπορούμε να δώσουμε και μια νέα όθηση στην οικονομία ολόκληρη. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να προσφέρει νομική ασφάλεια, προβλεψιμότητα, ε, μακροπρόθεσμα και ε, καινοτομία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να διευκολύνονται όσο και να ενθαρρύνονται. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και ελκυστική αγορά για δευτερογενείς πρωτεσίλες. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τους δείκτες, έχουμε κάνει ένα εργαστήριο εδώ στην Επιτροπή μας που έδειξε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία επιτάπητος ήδη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα το στόχο. Δηλαδή να είναι πάντα ξεκάθαρα τα δεδομένα και συγκρίσιμα. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να είναι και εφαρμόσιμοι και το διοικητικό ε, άθος να μην ανατινάξει όλο το πλαίσιο. Έχω κάνει σχετικά και προσωπικά μια τροπολογία. 30% έχουμε ε, θέσει ως στόχο για το 2030, αλλά εγώ με μια άλλη τροπολογία ε, τονίζει τη σημασία που έχει ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν το τρίτο. Τέταρτο, θέλω να έχουμε μια πολιτική για τα υλικά και για τα προϊόντα με πάρα πολύ σκέψη και περισυλλογή που να λαμβάνει υπόψη όλο το βίο ε, και τον κύκλο ζωής και τον οικολογικό σχεδιασμό και την αντίστοιχη νομοθεσία. Ο αντίκτυπος κάθε ε, νομοθεσίας βεβαίως θα πρέπει να εξετάζεται πολύ σωστά. Και πέντε για το πακέτο των αποβλήτων, τελευταίο. Και εδώ σας παραπέμπω σε μια τροπολογία μου και ένα δελτίο τύπου που έβγαλα μαζί με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές πρόσφατα ε, για τα απόβλητα. Ε, στόχοι πρέπει να είναι φιλόδοξοι με στήριξη αναχώρα, ειδική, ε, σαφούς ορισμούς, ε, εναρμονισμένες μεθόδους μέτρησης, σεβασμό για την ιεραρχία των αποβλήτων και ελάχιστες απαιτήσει για την ευθύνη των παραγωγών και των κατασκευαστών. Για μένα αυτό είναι ένα πλαίσιο απαραίτητο. Προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπολείπους και όλους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκερμπράντη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Σύρπα Πιετικάινεν για την εξαιρετική της έκθεση στο σχέδιο. Και ο Μάρκ Ντεμέσμακερ έχει απολύτως δίκιο ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ και έντονα για την κυκλική οικονομία. Για μένα αυτό δεν είναι έκπληξη. Είναι λίγα τα θέματα όπου η οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον πηγαίνουν τόσο πολύ ε, μαζί, χέρι-χέρι, όσο στην περίπτωση αυτή της κυκλικής οικονομίας. Αν κοιτάξετε την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο των αποβλήτων και την αντίστοιχη ανακοίνωση, θα διαπιστώσετε πόσο μεγάλη σημασία έχει πραγματικά η οικονομική πτυχή ε, είναι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Θα ε, σας δώσω μερικά αριθμητικά στοιχεία ε, της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ίδιας. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ετησίως μπορούν να εξοικονομούν πάνω από 600 δις ευρώ και μόνο αν μεταβούν σε αυτή την κυκλική οικονομία. Αυτό θα προσφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία μία όθηση 3,9% του ΑΕΠ. Αυτά είναι αστρονομικά νούμερα σε καιρούς όπου αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στο 1% της μεγέθυνσης της οικονομίας. Ε, ωστόσο, παρόλα αυτά, οι περισσότεροι θεωρούν αυτό το θέμα περιβαλλοντικό, που είναι μεν και περιβαλλοντικό, αλλά ε, ε, το περιβαλλοντικό είναι αυτό που μένει δωρεάν μετά από τα τεράστια οικονομικά ωφέλη. Και δείχνει πόσο περίεργο είναι ταυτόχρονα το γεγονός ότι η Επιτροπή Juncker αποφάσισε να αποσύρει το μόνο νομοθετικό πακέτο ε, αυτού του θέματος, το, τη δέσμη για τα απόβλητα. Αν δείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, παράγουμε μόνο 30% των πόρων που χρησιμοποιούμε. Άρα έχουμε τεράστια εξάρτηση από την εισαγωγή από τρίτες χώρες πρώτες ύλες και μεγάλη εξάρτηση, επαναλαμβάνω. Ρωτήστε οποιαδήποτε εταιρεία χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν είναι το υψηλό κόστος των πόρων. Αυτό είναι πρόκληση, αλλά το αντιμετωπίζουν οι εταιρείε. Το πρόβλημα είναι οι τεράστιες διακοιμάσεις των τιμών. Είτε είναι ξέρω εγώ, βιολογικές πρωτεσίλες ή άλλα υλικά. Οι διακοιμάσεις των τιμών είναι κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ τις εταιρείε και είναι από τους μεγαλύτερους εφιάλτες για κάθε εταιρεία. Αυτό μπορούμε να το λύσουμε προχωρώντας προς αυτή την κυκλική οικονομία. Λοιπόν, έχει σημασία όχι μόνο περιβαλλοντική και οικονομική τεράστια. Μερικά σχόλια για την εξαιρετική έκθεση της ΣΥΡΠΑ πιετικά είναι. Η δική μου πολιτική ομάδα πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα οικονομικά εργαλεία πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή αγορά για δευτερογενή υλικά. Με διάφορους τρόπους γίνεται αυτό. Με μετατόπιση της φορολόγησης, δηλαδή να μην φορολογείται η εργασία, οι πρώτες ύλες. Και με το ΦΠΑ μπορούμε να το δούμε για δευτερογενή υλικά. Κάποια στοιχεία που μπορούμε να δημιουργήσουμε αγορά για αυτά τα ε, υλικά. Και κάτι άλλο που έχω προτείνει στη δική μου έκθεση για την αποτελεσματική χρήση πόρων πριν από λίγα χρόνια, να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά αποβλήτων, ένα σέγγεν για τα απόβλητα, για χώρες που έχουν αρκετό τρόπο και σωστό διαχείριση των αποβλήτων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν εντό εισαγωγικών και απόβλητα από άλλε χώρε για να τα επεξεργάζονται. Αυτά, Πρόεδρε, δεν θέλω να επαναλάβω τα πολύ ωραία και σωστά που λέει η έκθεση για τον οικολογικό σχεδιασμό και άλλα στοιχεία. Κάτι άλλο σημαντικό επίσης είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στην αποτελεσματική χρήση ε, των πόρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως φέτος το έχει κάνει στην άκρη. Αυτό το έχει εξαιρέσει από την έκθεσή της. Και τέλος, Πρόεδρε, Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να επικεντρωνόμαστε σε κάποιες γραμμές του προεπολογισμού και ας πούμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων του Juncker για την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Δεν είναι όμως μόνο αυτό σημαντικό. Θα πρέπει να κοιτάμε και τον υπόλοιπο προπολογισμό και τις μελλοντικέ επενδύσεις του Ταμείου αυτού, στρατηγικών επενδύσεων, να μην πηγαίνουν ε, στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της κυκλικής οικονομίας. Να έχουμε πολύ περισσότερη συνοχή λοιπόν στην πολιτική μας. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και βλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί της και τους υπόλοιπους σκιώδες ηγητές. Ευχαριστώ. Κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα που ανέβαλε, ανέλαβε γιατί έπρεπε να υπόψη και τα δικά μας σχόλια, αλλά και τα σχόλια των διαφόρων κρατών μελών που είναι τελείως διαφορετικά τα συμφέροντά του, Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρεθεί κοινό έδαφος. Να πω ξεκάθαρα ότι οι στόχοι που θέτουμε πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να βασίζονται σε επιστημονικές αναλύσεις. Θα πρέπει να είναι εφικτοί και υλοποιήσιμοι στόχοι αυτοί. Κατά την άποψή μου, ο στόχος το 70% για την ανακύκλωση είναι υψηλό και πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Επίσης, θα έπρεπε να είναι και πιο φιλόδοξη η Κομισιόν στις προτάσεις της σε κάποιους άλλους τομείς πέραν της ανακύκλωσης. Παραδείγματο χάρη. Καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν όχι μόνο τα δημοτικά απόβλητα, αλλά και τα εμπορικά και βιομηχανικά. Δεν πρέπει να παρεξηγήσετε, γιατί ο περιορισμό των αποβλήτων σίγουρα είναι κάτι αποφελέ και η ανακύκλωση ίσως να είναι ε, ο βασικός τρόπος για μια αηφόρη οικονομία. Όμως, είναι σημαντική και η διατύπωση ε, των στόχων Καλά να τα γράφουμε αυτά, αλλά πρέπει και οι στόχοι που θέτουμε να είναι ρεαλιστικοί. Σε ό,τι αφορά την ε, υποχρεωτική διαλογή των ε, αποβλήτων είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνη. Για την παραγωγή ενέργεια επίση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα. Είναι μια ιδέα που ξέρω ότι δεν βρίσκει σύμφωνο πολλού συναδέλφου. Πρέπει να είμαστε όμω ρεαλιστέ. Κάποιοι θα ήθελαν, κάποιοι ιδεαλιστές, μια ε, εντελώς απαλλαγμένη από, απόβλητα κυκλική οικονομία, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε ε, το τέλειο ε, σε επίπεδο 100%. Οι επιστημονικές γνώσεις και οι προσεγγίσεις των κρατών μελών δεν μας επιτρέπουν να ελπίσουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη τέλεια οικονομία 100%. Βέβαια δεν πρέπει να κάψουμε μαζί με τα ξέρα και τα χλωρά. Βέβαια, η διαλογή είναι ένα σημαντικό θέμα και η ανακύκλωση. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα απόδειτα για να αντικαταστήσουν ενδεχομένω κάποιους πρωτογενεί πόρου που χρησιμοποιούμε τώρα. Βέβαια, η καύση αποβλήτων είναι κάτι που δεν θα μας επιτρέπει ταυτόχρονα να παραγαγούμε ενέργεια, θα έπρεπε να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Τώρα, διατροφικά απόβλητα, προβληματική προσέγγιση. Και αυτό δεν θα αλλάξει αν δεν ορίσουμε σωστά τα διατροφικά απόβλητα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Έχουμε τα βιολογικά απόβλητα. Τώρα το να λέμε αν είναι φυτικά ζωικά και αν είναι τρόφιμα ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Έχω καταθέσει τροπολογίες με στόχο να γίνουν κάποιες διορθώσεις ε, και βελτιώσεις τα δομικά απόβλητα από την ανακαίνιση κτηρίων ε, ή την ανέγερση κτηρίων. Ποιοι είναι οι στόχοι για το 2025 και το 2050 για τα δομικά απόβλητα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Πάντως οι τροπολογίες μου στόχο έχουν να απευθύνω μια έκκληση στην Κομισιόν την οποία καλώ να δει ποιες είναι οι οικονομικές δομές των αμονωμένων κρατών μελών και ποιες είναι οι ανάγκες τους. Τέλος. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι πολύ συχνά παραπονούμεθα για την κακή ποιότητα της νομοθεσίας. Δυστυχώς όμως τα ίδια λάθη που, για τα οποία παραπονούμεθα, στα ίδια αυτά λάθη υποπίπτουμε και εμείς. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να ορίσει καλά τι εννοεί απόβλητα και τι εννοεί απόβλητα ως πόρο. και χρησιμοποιείται και κάποια άλλη ορολογία για τους πόρους, την οποία επίσης θα πρέπει να την διευθυνήσει ακόμη περισσότερο η Κομισιόν. Και τα απόβλητα πρέπει να οριστούν καλύτερα και η προσέγγιση θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέψει τη μετρίαση του διοικητικού φόρτου. Πρέπει να είναι σαφές αυτά που λέμε, να είναι εύληπτα, κατανοητά πρέπει να ορίσουμε και να διασαφηνίσουμε κάποιους όρους του κειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε καμιά εναρμόνιση και ούτε βέβαια θα πετύχουμε τους στόχους μας και τις φιλοδοξίες μας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λέω κύριο Σέικχαουτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να στείλω συγγνώμη εκ του κυρίου Τούρμες, ε, τον οποίο αντικαθιστώ γιατί δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Είναι ένα θέμα βέβαια που με ενδιαφέρει, οπότε δεν με πειράζει καθόλου, που δεν είναι εδώ ο κύριος Τούρνος. Αλλά αυτό να μην του το πείτε βέβαια. Καταρχά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω θερμά την φίλτρα κυρία Πίτη Κάινεν για τη μέχρι τώρα εξαιρετική τη δουλειά και για τι τροπολογίε θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου. Ξέραμε ότι έχουμε ένα περιορισμό ε, με τη, στο, ως προς το περιεχόμενο, αλλά με τις τροπολογίες νομίζω ότι πλέον μπορούμε να ξεδιπλώσουμε πιο πολύ τη θέση μας απέναντι στη θέση της Κομισιόν που εξεργάζεται από ό,τι μας λένε και μια πιο φιλόδοξη πρόταση τώρα. Θα ήθελα πάντως και την Κομισιόν να την ευχαριστήσω. γιατί τελικά αυτό το θέμα προσέλκυσε τη μεγάλη προσοχή όταν το πορό ακούστηκαν αυτέ οι φήμες ότι ίσως να ανακαλέσει την πρόταση, την θετική πρόταση η Κομισιόν και εγώ είχα προσπαθήσει να εξηγήσω στου δημοσιογράφου, τι συμβαίνει. Πολλοί δημοσιογράφοι τότε μου είπαν ναι, η κυκλική οικονομία ούτε και ξέρω τι περί πρόκειται, αλλά τέλος πάντων, ε, ήδη εμείς εδώ και καιρό μιλάμε για αυτή την κυκλική οικονομία, αλλά έξω ο κόσμο ε, δεν αντιλαμβάνεται ευθύ αμέσω περί πρόκειται. Άρα, με αυτή την έννοια, η κυκλική οικονομία ήταν δύσκολο να μπει και στι εφημερίδε ω θέμα, αλλά χάρη στην Κομισιόν πρέπει να πω ότι ακόμη και οι μεγάλε εφημερίδε μιλάνε για την κυκλική οικονομία πλέον. Άρα, από αυτήν την έννοια, μάλλον τη αξίζει τη Κομισιόν ένα ευχαριστώ γιατί έριξε προβολή στη δημοσιότητα στην κυκλική οικονομία με την απειλή τη απόρριψη, τη απόσυρση αυτή τη πρόταση. Και τώρα έχω μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Είναι σημαντικό βέβαια να πούμε και εμεί ε, ω Κοινοβούλιο τι περιμένουμε από μια τέτοια πιο φιλόδοξη πρόταση από την Κομισιόν. Και γι' αυτό θα πρέπει και η Κομισιόν να παρακολουθεί του σύνεγγυ στη δική μα δουλειά εδώ. Έρχομαι στο περιεχόμενο μου αρέσει και το έκανα και για ποιητικά είναι να δει το ανάρτη και κατάντη, upstream dance, Όχι μόνο την ομψία περί αποβλήτων, αλλά και τι πρέπει να γίνει ανάντι. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, η πλήρη εφαρμογή τη συστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα σίγουρα είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Επίση, πρέπει να μα απασχολήσει η πρόληψη, η μείωση και η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Αυτά τα θέματα είναι κρίσιμα και μετά έχουμε και τους στόχους ανακύκλωσης που εντάσσονται στις μετρητά για τα απόβλητα. Θα χρειαζόμαστε όλα αυτά μέτρα. Τώρα, σε σχέση με τη Σάφο Κονέτσνα που μίλησε για την καύση των αποβλήτων, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι εμεί δεν θέλουμε την καύση ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ε, αν απαγορεύουμε σχοματερές και θέλουμε να υπάρξει ανακύκλωση, τι θα γίνει. Τελικά θα καίγονται τα πάντα. Το βλέπουμε ήδη, ε, υπάρχει αποτέφρωση σε πάρα πολλές ε, ε, χώρες. Και αντί να βλέπουμε, αντί της ε, να αυξάνεται η ανακύκλωση, βλέπουμε να αυξάνεται η αποτέφρωση. Και είμαστε και στη, και στη χώρα μου αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο πλέον ειδικοί σε αυτό. Το θέμα είναι να μην καίμε τα ανακυκλώσιμα απόβλητα. Τώρα, ανάντι. Πρέπει να πω ότι ο οικολογικός σχεδιασμός είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, αλλά και η υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών. Η κυρία να το είπε νομίζω, ότι ναι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όμως είναι σημαντικό να φροντίσουμε, γιατί πράγματι αν θέλουμε επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, πρέπει να μην περιλαμβάνουν ουσίες που θέλουμε να κυκλώσουμε ή να ξαναχρησιμοποιήσουμε, να μην περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες. Και πολλές ε, εταιρείε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συζήτηση περί κυκλικής οικονομίας ε, για να μειώσουν ε, τα πρότυπα της νομοθεσίας REACH. Είναι σαν χόμπι για μερικούς. Δεν νομίζω όμως ότι η κυκλική οικονομία σημαίνει ότι είναι πολύ περιοριστική νομοθεσία REACH. Όχι, αντιθέτως δεν πρέπει οι επικίνδυνες ουσίες ε, να ε, μπαίνουν καν στην ε, διαδικασία της ανακύκλωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Και έρχομαι σε μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Σκερπράντη για την ιδέα αυτή για το Σέγγεν. Σας θαυμάζω που επιμένετε τόσο πολύ σε αυτό το θέμα. Ήδη στο σχέδιο έκθεσή σας για την ε, ενεργειακή, για την αποδοτική χρήση των πόρων ε, το είχατε, αλλά τώρα επειδή αυτό και προσπάτα να το περάσετε πάλι από την πίσω πορτά. Δεν θέλουμε όμως εμείς αυτό να συμβεί. Και θα επιμείνω και εγώ από την πλευρά μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πιεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, προσυπογράφω κάθε λέξη του συναδέλφου Άικχαουτ όταν αναφέρθηκε στα όσα είπε η συνάδελφος Κονέτστα και εμείς συμφωνούμε ότι η αποτέφρεση ε, τα καίει όλα. Δεν υπάρχει μια ενδιάμεση φάση να διασωθούν κάποια απόβλητα. Και ξέρουμε ε, τελικά από καταλήγει η αποτέφρωση και τι συνέπειες έχει. Τώρα, εμείς ήδη από την αρχή είχαμε τη θέση της μείωσης της παραγωγής των αποβλήτων. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε για μια κυκλική οικονομία όσο γίνεται λιγότερη κατανάλωση ορυκτών πόρων. Για να είναι αηφόρος η οικονομία και βιώσιμα θα πρέπει να ε, αρχίσουμε να ε, απομακρύνουμε και να αποκλείουμε οτιδήποτε βλάπτει το περιβάλλον, τα ορυκτά και τα λοιπά. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή ε, και δεν θα πρέπει να... Ε, ε, βέβαια δεν μου αρέσει να μιλάω για την Ιταλία, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε κρατικές ενισχύσεις ή άλλες ενισχύσεις σε ορυκτές πηγές. Εμείς στην Ιταλία δίνουμε 6 δισεκατομμύρια το χρόνο για να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το 10% μόνο πάει στις ανακυκλώσιμες πηγές. Αιωλική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, ε, ηλιακή κτλ. Τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην ενίσχυση της αποτέφρωσης και το 50% για να δώσουμε ε, ενθάρρυνση και κίνητρα ε, στο πετρέλαιο, λες και είναι ανακυκλώσιμη και φόρος ε, πηγή ενέργεια. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε, να εκτοπίσουμε και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για κυκλική οικονομία. Σωστά τα λέει η συγκήτρια γιατί ε, δίνεται κίνητρο, ας πούμε, μείωση του ΦΠΑ για την ανακύκλωση και φορολογικά κίνητρα άλλα όταν χρησιμοποιούν εταιρείε ανακυκλωμένα υλικά και εκείνος που ε, παράγει με λιγότερους πόρους, ε, υπάρχει και μικρότερη κατανάλωση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πιστοποιητικό και ένας στόχος ξεχωριστός για την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών για να μειωθεί η παραγωγή των ε, αποβλήτων. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό και οικονομικό το 1 τρίτο των ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων που δεν πηγαίνουν στις χωματερές ε, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και δημιουργούνται και θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας φιλόδοξος στόχος ανακύκλωσης. Είναι δυνατό αυτό. Εμείς δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε και με τη συνάδελφο Κονέτσινα ότι θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξους αλλά και ρεαλιστικούς στόχους. Αλλά η πρόταση της ηγήτριας για το 70% μας βρίσκει σύμφωνος. Θα θέλουμε στα αστικά απόβλητα μέχρι το 2025 να ε, απαγορευτεί η αποτέφρωσή τους και κάθε είδους απόβλητο μέχρι το 2030 και να όπως σας είπα και στην ε, πρόταση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου συμφωνούμε ότι οι οικοδομές και οι κατασκευές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανακύκλωση και στην κυκλική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη και να εθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ανακαινίζουν τα κτίρια. Θα πρέπει να ε, προτιμούμε ε, μεθόδους κατασκευών που να επαναχρησιμοποιούν υλικά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στα κτίρια. Είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια και τους κοιόδους εισηγητές για να ε, έχει την τελική, όσο γίνεται καλύτερη μορφή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε. Να συνεχίσουμε αν θέλει και άλλος συνάδελφος να μιλήσει. Ε, θα πρέπει μέχρι τις 5.30 να έχουμε τελειώσει γιατί έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γεωργίας για την κλεονοποίηση. Ε, παρακαλώ λοιπόν όλα τα μέλη να ε, μειούν λίγο, το πολύ δυόμιση λεπτά, θα το προτίμηση δύο, η κυρία Γκροστέ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη συνάδελφα μας κυρία Πιετικάινεν για το έργο της και βέβαια η κυκλική οικονομία σήμερα είναι ένα ουσιαστικότατο θέμα, γιατί είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Γίνεται λόγος για ενεργειακή μετάβαση. Εγώ θα έλεγα και ότι η οικονομία μας θα πρέπει να δελθεί μια μετάβαση για να περάσει προς μια κυκλική οικονομία με επιτάχυνση και με πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους που έχουν τεθεί στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι στόχοι που αφορούν την ανάπτυξη ε, και την απασχόληση είναι στη στρατηγική 2020. Όταν γίνεται λόγος για όγκους αποβλήτων και τα λοιπά, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εναρμονίσουμε τις μεθόδους μέτρησης για να καταλήγουμε σε στατιστικές που να ε, πιστοποιούν και να περιγράφουν πιστά την πραγματικότητα. Υπάρχουν τα αστικά απόβλητα, δεν αντιλέγω, αλλά θα πρέπει κυρίως να επιμείνουμε ε, στην ε, ανακύκλωση και στη διαχείριση των εμπορικών και βιομηχανικών μη επικινδύνων αποβλήτων. Και πολλές φορές ε, η ανάκτησή τους είναι και πιο χρήσιμη γιατί είναι καλύτερης ποιότητας. Γίνεται λόγος για κυκλική οικονομία. Δεν σταματήσουν οι χωματερές, δεν διαφωνώ καθόλου. Να σταματήσει και η αποτέφρωση. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχεις ένα προϊόν που έχει γίνει απόβλητο και θα ανακυκλωθεί ή θα επαναχρησιμοποιηθεί μία φορά, δυο, τρεις φορές, μετά την τρίτη χρήση ε, είναι σκουπίδι. Δεν μπορεί πια ούτε να ανακτηθεί ούτε να ε, ε, επαναχρησιμοποιηθεί, να ανακυκλωθεί. Μπορεί λοιπόν στην τελική φάση αυτή να χρειάζεται κάποια αποτέφρωση. Ε, εκεί είναι η δυσκολία. θα πρέπει οι μονάδες αποτέφρωσης να μην είναι γιγαντιαίων διαστάσεων όπως ισχύει συχνά σήμερα για να μην ενθαρρύνουν στην αποτέφρωση. Η αποτέφρωση θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση όταν όλα τα άλλα έχουν εξαντληθεί. Και δεν μπορεί να παραταθεί άλλο ο βίος ενός προϊόντος που είναι πλέον οριστικό απόβλητο. Και όταν ε, γίνεται λόγος για ε, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική ε, αυτή η κυκλική οικονομία. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες Πάντω υποστηρίζω απολύτως την έκθεση της κυρίας Πιετικά είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριος Γκρότε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να απευθυνθώ στην εισηγήτρια και να την ευχαριστήσω διότι εδώ έχουμε πραγματικά τη συμμαχία των προθήμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ακούσουμε όλα αυτά που λένε οι συνάδελφοι και να μετρήσουμε πόσοι μίλησαν, ε, κάτι καλό θα βγάλουμε και ε, θα πρέπει να πιέσουμε κάπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού εδώ επικρατεί τόσο μεγάλη ε, συνένεση και σύμνοια. Και τουλάχιστον έτσι στα ρετυρέ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα μεγαλύτερο θάρρος και περισσότερο ε, ε, ε, όταν βλέπουμε τη μοίρα επιφυλάσσουν το πακέτο ε, των αποβλήτων. Δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, θέσεις εργασίας θα ε, δημιουργηθούν αν το εφαρμόσουμε σωστά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε. Υπάρχει αυτό το δυναμικό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί δεν έχουμε ε, τόσο πολλές βιώσιμες και καλές θέσεις εργασίας για να είμαστε τόσο επιπόλαιοι με αυτό το θέμα και επιφανειακοί. Μερικά σημεία και τροπολογίες δικές μου θέλω να αναφέρω πρώτον. Ε, η σπατάλη τροφίμων. Θα πρέπει να συνηθίσουμε στο μέλλον σε όλες τις εκθέσεις, είτε είναι στη γεωργία είτε είναι εδώ στο περιβάλλον. Όταν πρόκειται για ασφάλεια τροφίμων θα πρέπει να κοιτάμε τι επιπτώσεις έχει η νομοθεσία μας ως προς τη σπατάλη τροφίμων. Θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποιοι δείκτες έτσι ώστε να ξέρουμε, να μετράμε με ένα σύστημα δικτών ε, τι συνέπειες θα έχει η απόφασή μας στη σπατάλη των τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε ποιο βαθμό μπορούμε ε, να προωθήσουμε κάποια πράγματα, όπως το leasing, δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα πολλές φορές ή το car sharing που να μοιραζόμαστε ένα αυτοκίνητο ε, και αυτή η κυκλική οικονομία πώς μπορεί να διεισδύσει στη ζωή του καθενός και να ε, το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και μια παράκληση, τώρα που είναι αρχή. Όταν έχουμε καλές διαδικασίες για την ανακύκλωση των αποβλήτων και έχω υπόψη μου στην εκλογή μου περιφέρεια μια περίπτωση όπου ε, υπάρχει υγρή ε, ζύμωση και στεγνή ζύμωση η μία πάνω στην άλλη. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι αυτά ε, τα στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να παραμένουν σε χωματερές. Ε, το ξέρω ότι πάντα υπάρχουν κατάλοιπα, τη φυσική τι να κάνουμε, δεν μπορείς να την καταργήσεις. Ε, βλέπω το σφυράκι ήδη, παρακαλώ να τα λάβετε αυτά υπόψη, να προσέξουμε, να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά και πριν ξανακούσω κανένα σφυρί σταματάω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, να συγχαρώ τη συνάδελφο για αυτή την έκθεση που είναι εξαιρετική βάση εργασία. Περιμένουμε με ανυπομονησία τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά και την έκθεση αυτή. Θέλουμε με αφορμή την έκθεση να εκφραστούμε σε ένα θέμα κεφαλαίου σημασία για το μέλλον τη Υπήρου. Ήθελα να δώσω έμφαση σε κάποια σημεία μόνο. Πρώτον, αυτό που αναφέρει και ο συνάδελφο Γκροστέτ Εναρμόνιση. Εναρμόνιση των στατιστικών μεθόδων. Πρέπει να υπάρξει τέτοια εναρμόνιση ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί από τη σκοπιά της κυκλικής οικονομίας. Δεύτερον, η εδαφικότητα. Η κυκλική οικονομία θα πρέπει να οριστεί ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών με, τον, με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρξει προμήθεια σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά με βάση τις τοπικές ανάγκες ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις στον ανεφοδιασμό. Θα ήθελα επίσης να επικεντρωθώ στην διασπάθηση των τροφίμων, την κατασπατάληση τροφίμων. Εδώ είμαστε υπεύθυνοι για το θέμα αυτό στη Γαλλία. Εγκρίναμε νόμο για, κατά της κατασπατάλησης των τροφίμων και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε στο τι ορίζεται ως ε, διασπάθηση και κατασπατάληση τροφίμων. Γι' αυτό συμφωνώ με την τροπολογία 343 και για να ολοκληρώσω, μια και πρέπει να είμαστε συνοπτικοί πρόεδρε, να πω ότι θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτή η αρχή πρέπει να οριστεί και οι τροπολογίες 66, 160 και 161 που αντίκεινται στην αρχή αυτή δεν με βρίσκουν συμφώνη. Ευχαριστούμε κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη σαφή και περιεκτική έκθεση και σημειώνω και εγώ ότι πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες έχουν υποβληθεί. Δείχνει αυτό πόσοι ε, σημασία δίνουμε όλοι στην ε, συγκεκριμένη έκθεση και στην δέσμη μέτρων που αποσύρθηκε για τα απόβλητα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο, ένα νέο μοντέλο. Αυτό της κυκλικής οικονομίας. Αλλά όχι μόνον για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία είναι καθοριστική σημασία, αλλά και για άλλους λόγους, όπως αυτούς που ανέφερε ο συνάδελφος και ο συνάδελφος Γερμπράντη. Δηλαδή θέλουμε αυτός να γίνει ένας από τους άξονες της ανάπτυξής μας και της οικονομικής και της ανταφικής. Το 40% του κόστους πρώτων μελών για μια επιχείρηση, ένα από τα δεδομένα που μα έδωσε η συγκέντρια στην έκθεση, είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά μας και το δίκτυο των επιχειρήσεων που δημιουργούμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων είναι βασικό στοιχείο για να ξεκινήσουμε στην οποιαδήποτε προσπάθεια ανάπτυξη και όσα θέλουμε να κάνουμε για την κυκλική οικονομία. Εάν θέλουμε να δέψουμε ταχαίω λοιπόν προ την κυκλική οικονομία, πρέπει να εντοπίσουμε τομεί τη ευρωπαϊκή οικονομία που ακόμη έχουν σημαντικά, ε, σημαντικά οικονομικά εμπόδια προτού ενταχθούν στην κυκλική οικονομία. Γι' αυτό υποβάλαμε και εμεί κάποιε τροπολογίε μαζί με του υπόλοιπου συναδέλφου και είναι και τρει οι φάσει στι οποίε θέλουμε περισσότερο να επικεντρωθούμε. Πρώτα απ' όλα, την, τον βιώσιμο σχεδιασμό των προϊόντων, κάτι που το έχει αναπτύξει αρκετά η η κατανάλωση. Θα πρέπει να προγραμματίζουμε το πώ ε, θα σχεδιάζονται τα προϊόντα αλλά και τα κατάλληλα που θα αφήνουν, κάτι που έχει να κάνει με την κατανάλωση, αλλά εγώ περισσότερο θα επικεντρωνόμουν στον σχεδιασμό. Και μετά και ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Διότι αν θέλουμε να ανακτήσουμε πρωτεσίλε θα πρέπει να δράσουμε προφανώ. Ε, εντάχει, νομίζω ότι κεντρικό σημείο είναι συμβατή, ο συμβατό σχεδιασμό για να ορίσουμε πόσου και ποιου πόρου μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε, τη στιγμή όμω ήδη που συλλαμβάνουμε τα προϊόντα. Στην επόμενη λοιπόν οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την νομοθεσία μόνο ο σχεδιασμό των ενεργειακών αλλά δεν έχουν οριστεί υποχρεωτικά κριτήρια ως προς την ανακύκλωση, την ε, επαναχρησιμοποίηση και την αξιοποίηση. Σε ό,τι αφορά το μέρος της ανακύκλωσης και της ανάκτησης, εδώ αναμφίβολα θα πρέπει να ορίσουμε δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με αυτούς που τώρα ισχύουν και που δεν θα πρέπει να είναι κατώτεροι από την πρόταση που είχε υποβληθεί προκαιρού και αποσύρθηκε. Θα πρέπει να υπάρξει ένας μια εναρμονισμένη μεθόδος υπολογισμού για να μπορούν να γίνονται και συγκρίσει και δεν θα μπω στην ουσία τη καύση ή τη αποτέφρωση που έχει προκαλέσει τεράστιε συζητήσει ε, για το τι θα γίνεται ακριβώ με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Όμω ε, θα πρέπει να δούμε την ενεργειακή, την ενεργειακή ανάκτηση σε περίπτωση με κεκλώσιμο υλικών. Και κάτι ακόμη που είναι σημαντικό, να αποφύγουμε τις ε, διαρκείς εξαιρέσεις εκεί που τα κράτη δεν μπορούν κάποια στιγμή να εφαρμόσουν τις διατάξεις. Αν θέλουμε κυκλική οικονομία, αυτό είναι ένα βασικό σημείο αφετηρίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Σχέιο Πύρικ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Πιετικά, είναι πάρα πολύ ωραία έκθεση. Έχω κάνει κάποιες τροπολογίες. Ε, εγώ εργάστηκα στην Ολλανδική Βουλή σε αυτά τα θέματα πάρα πολλά χρόνια και ε, είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες αυτό με τα απόβλητα. Ε, θα πρέπει ε, οι τροπολογίες μας να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και να έχουν να κάνουν με την υλοποίηση και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Εάν γίνει αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη θα έχουμε προχωρήσει πολύ. Δεύτερο, να απαγορευτούν οι χωματερές, να το κλείσουν. Ε, η χώρα μου δεν το κάνει αυτό, άλλες χώρες το κάνουν, ε, αλλά το σημαντικότερο είναι ε, να γίνεται η διαλογή των αποβλήτων, να υπάρχουν συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν και υπάρχουν στην Ολλανδία, στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε, να τις αξιοποιούμε. Έχουμε λεφτά για τα διάφορα ταμεία, το παιδιωτικό ταμείο, όλοι χτυπούν την πόρτα για να κάνουν κάτι με τα απόβλητα, ας τους αφήσουμε. Και τέλος ε, για την αποτέφρωση. Η συνάδελφος Γκροστέτ μίλησε για τις ε, εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Συμφωνώ με τα όσα λέει, αλλά εγώ ζω ε, στην ε, Ολλανδία, στο Τβέντε και τι γίνεται. Ε, χρειαζόμαστε δέντρα για να λειτουργούν αυτές οι εγκαταστάσεις και κόβουν τα δέντρα μας και αποψηλώνονται το δάσος για να λειτουργήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλέκ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τώρα θα συνεχίσω στα κρατικά. Θέλω να je ovdje bilo nekoliko puta spomenuto i problem spaljivanja otpada. Πολλές φορές μιλήσαμε για αποτέφρωση αποβλήτων και για κυκλική οικονομία. Στην κυκλική οικονομία η αρχή της καύσης των αποβλήτων Είναι κάτι που θεωρείται απαραίτητο, αλλά το θέμα είναι να επενδύσουμε ως το δυνατόν περισσότερο στη γνώση για την ε, ιεράρχηση των αποβλήτων. Το θέμα είναι και ο σχεδιασμός των προϊόντων που είναι χρήσιμα για την κυκλική οικονομία. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει προτάσει στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ζωή, ε, ηλεκτρονικό εξοπλισμό κτλ. Διότι έχουμε τις υποψίες ότι μειώνουν οι κατασκευαστέ ε, σκοπίμως τη διάρκεια ζωής αυτών των ε, ειδών εξοπλισμού για να αντικαθίστανται πιο γρήγορα. Εμείς όμως θέλουμε να αποφεύγουμε, αποφεύγουμε τα απόβλητα λογική καινοτομία και κολλικό ε, σχεδιασμό πρέπει να δημιουργούν ε, νέα προϊόντα, νέε συσκευασίε με στόχο και τη μείωση του κόστου. που μπορεί να προέλθει από την αγορά νέων συσκευών. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε επίσης τη συσκευασία των προϊόντων αυτών να την ξαναχρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς και μετά να ανατυπλώσουμε αυτή τη συσκευασία ή να την διαθέσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Nano. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ενανό, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Πιτικανέν για την εκθεσή της, για την όλη έννοια της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να προβλέψουμε και την τοπική διάσταση. Για αυτό το σκοπό δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις εθνικές στρατηγικές προκειμένου να μειώσουμε το, την ε, έκταση των ε, δικτύων. Διότι όσο είναι μεγαλύτερε οι αποστάσει, τόσο περισσότερα εμπόδια θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι αντιευρωπαϊκές απόψεις που αναπτύσσονται εδώ είναι ένα παράδοξο στην ε, εξέταση του Θα ήταν προτιμότερο έμφαση να δώσουμε σε στόχους ρεαλιστικούς, δηλαδή όχι το 0% αποβλήτων ε, και κυρίως να κοιτάξουμε τα τοπικά δίκτυα και τις τοπικές οικονομίες. Ε, νομίζω μεριμνά μας θα πρέπει να είναι να δώσουμε συστάσεις για επί της ουσίας πραγματικές ε, διαδικασίες που πρέπει να αναπτυχθούν και όχι για υπερφιλόδοξους, υπερκρατικούς στόχους. Με τα απορρίμματα θα πρέπει να περιορίσουμε και την ανεξέλεγκτη, ε, τις ανεξέλεγκτες ελεύθερες συναλλαγές που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα. Ευχαριστούμε ο κύριος Ζιγκζιμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ υπάρχουν κάποιες πτυχές που ανέπτυξε η κυρία Πετικάινεν στην έκθεσή της για την οποία θέλω να την συγχαρώ διότι κάποιες από αυτές τις πτυχές είναι πολύ σημαντικές και θέλω να τις αναπτύξω τώρα. Πρώτον, ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος. Το ανέφεραν ήδη κάποιοι. Οπωσδήποτε για κάποια καταναλωτικά αγαθά ισχύει. Ο κύκλος ζωής η θελημένα είναι πιο σύντομο, για να το πω έτσι. Ή τέλο πάντων υπολογίζεται προσεκτικά. Και θα πρέπει να ε, εξετάσουμε το κατά πόσον ισχύει ο κύκλο ζωή αυτό στην πραγματικότητα και θα πρέπει να υπάρξει μετά ε, αντικατάσταση. Απόσυρση του προϊόντο και αντικατάσταση με ένα νέο. Έτσι, πολλέ φορέ βέβαια έχουμε και υπέρμετρη, υπερητή κατανάλωση για κάποια προϊόντα που καθίστανται περιτά ενώ θα μπορούσαν να έχουν σχεδιαστεί απλώ καλύτερα. Δεύτερο σημείο. Τα συμβατικά απόβλητα είναι ένα στοιχείο, αλλά με τα οργανικά τι γίνεται. Το, ε, το 1989 παρήγαμε 80 εκατομμύρια τόνους οργανικών απορριμμάτων, ε, μεταξύ των οποίων τρόφιμα και μάλιστα επεξεργασμένα, τα οποία απλώ πετώνται, θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί. Να έχουν αξιοποιηθεί. Μιλάμε για τρόφιμα που ούτω ή άλλω δεν είχαν περάσει την ημερομηνία λήξη. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στον ανάγκη περιορισμού της κατασφατάλησης τροφίμων. Μιλάμε για τρόφιμα που κατασπαταλήθηκαν δεν καταναλώθηκαν. Δεν φαγώθηκαν ή πετάχτηκαν επειδή είχε περάσει η ημερομηνία η ημερομηνια ληξη τους. Είναι το ένα τρίτο των ε, απορριμμάτων των οικοκυριών αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ε, δεδομένης της του πληθυσμού παγκοσμίω. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός φτωχών ανθρώπων ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δεν, ε, τους οποίους δεν αφορά η ασφάλεια. 80 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων λοιπόν είναι ένα σωρό ενέργεια που θα μπορούσε να έχει εξοικονομηθεί ακόμα και αν ε, δεν ήταν για τρόφιμα που τελικά οδηγήθηκαν σε καύση. Δεν μπορούμε λοιπόν απλώς να πετάμε τα τρόφιμα. Now I ask Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μπόπελ. Έχετε τον λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Είναι χρήσιμες τροπολογίες. Ε, ε, προσθέσατε επίσης κάποιες αναφορές για περιβαλλοντικά επιζήμιες ουσίες ή τηρητή μνήμα στις νέες δεξιότητες που απαιτούνται, ΜΜΕ, έτοιμα η παραγωγή και τα, ε, τα τρόφιμα να από μια λογική πολιτική και αυτό σχετίζεται σίγουρα με τον οικολογικό σχεδιασμό. Η χρήση της βιομάζας πράγματι πρέπει να ε, εξεταστεί περισσότερο και στο πλαίσιο της ενέργειας που σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει σήμερα, αλλά και σε ό,τι αφορά εναλλακτικές χρήσεις ε, της βιώματος ως υλικού και της ε, όλης ε, βιωσιμότητας. Ε, η μέτρηση επίσης και σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για, τις δείκτες, για τους δείκτες. Ξέρετε ότι επεξεργαζόμαστε δείκτες για την κατανάλωση των πρώτων υλών. το είχαμε προτείνει να έχουμε έναν δείκτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται στα απόβλητα και να καλύπτει διάφορα υλικά ή ουσίες. Δεν μπορούμε με βάση αυτό όμως ακόμη να θέσουμε δεσμευτικούς στόχους. Έχουμε βέβαια την αποσύνδεση που θα μπορούσε να προκύψει λόγω του στόχου 30% μέχρι το 2030, για του 30% μείωση. Πάντως αυτοί οι δείκτες ναι μεν μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο, θα μπορούσαν να προκύψουν ε, ε, κάποια εμπορικά αντισταθμίσματα αν δεν σχεδιαστούν σωστά αυτοί οι δείκτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους για τα απόβλητα, απεξεργαζόμαστε και θα υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση για την θεώρηση των στόχων των αποβλήτων στο τελευταίο τρίμηνο του 2015. Και αυτό θα γίνει από κοινού και με τα άλλα στοιχεία της δέσμευσης μέτρων για την κυκλική οικονομία. Σίγουρα ε, θα ε, επιδιώξουμε τους στόχους του 7ου προγράμματος δράση για το περιβάλλον. Θέλουμε όμως να λάβουμε υπόψη μας και τις διαφορετικές αφετήρες και πραγματικότητες των κρατών μέλων. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μια δημόσια διαβούλευση ε, θα ξεκινήσει την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να ακούσουμε περισσότερα στοιχεία για άλλες πτυχές της κυκλικής οικονομίας που δεν αφορούν τα απόβλητα και θα γίνει και μία ε, διάσκεψη στις 25 Ιουνίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια. Βέβαια, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγα λεπτά πρέπει να αλλάξουμε αίθουσα, γιατί έχουμε την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΕΝΒΙΑΓΡΙ. Κυρία Πιετικάινεν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναντέλφους για τα πολύ καλά επικοδομητικά σχόλια. Νομίζω τα περισσότερα εύκολα θα τα συμπεριλάβω στην έκθεση και σίγουρα θα βελτιώσουν την ποιότητα της γνωμοδότησής μας σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Να πω επίσης ότι ότι η Γαλλία αξίζει συγχαρητηρίων που παγορεύει την κατασπατάληση των τροφίμων, τα τροφικά, διατροφικά απόβλητα. Να ένα καλό παράδειγμα τι μπορεί να πετύχει η νομοθεσία. Και βέβαια η δράση του κλάδου των τροφίμων ε, που είναι το ένα τρίτο των οικιακών αποβλήτων. Είχα ξεχάσει να μιλήσω για κάποιες τροπολογίες. Τέλος πάντων, το τελευταίο σημείο που νομίζω θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο είναι αυτό το ζήτημα μεταξύ ε, χωματερών έναντι ε, μονάδων αποτέφωσης. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε δείκτες. Γιατί πράγματι υπάρχουν απόβλητα που δεν μπορούν να συλλεγούν ε, με διαφορετικό τρόπο. Είναι κάποια απόβλητα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Και το μόνο που μένει είναι ή να αποτεφραθούν ή να διατεθούν οριστικά. Ποιο είναι όμως αυτό ε, το ποσοστό. 5% όλων όσων ε, πηγαίνουν στις, στις, ε, στους χώρους υγειονομικής ταφής. Τι κάνουμε. με αυτά τα απόβλητα τα οποία καταλήγουν ε, σε όπως τα λάστιχα τα οποία καταλήγουν ε, στην ε, μονάδα αποτεύρωσης γιατί δεν μπορεί να παραχθεί ενέργεια από την στις χωματέρες μάλλον γιατί δεν μπορεί να παραχθεί ενέργεια από την αυτούς και τα λοιπά. Επίσης έχουμε την ξεχωριστή διαλογή, έχουμε επιχειρηματικά μοντέλα. Εκεί από τη ροή των αποφτών βγαίνουν οι πρώτε ύλε. Και με συναδέλφου από την Πολωνία και άλλου Ανατολικοευρωπαίου έχω συζητήσει και μου είπαν ε, ότι υπάρχει και πρόβλημα ε, με την ευρεία αυτή εκτεταμένη αποτέφρωση. Υπάρχει θέμα κόστους. Γι' αυτό το σκέφτομαι κι εγώ. Και πρέπει να δούμε αν ε, υπάρχουν ή μπόρει να υπάρξουν πανευρωπαϊκές δομές για συγκεκριμένα απόβλητα. Εμείς θα έχουμε προβλήματα και στη Φιλανδία και θα υπάρχουν και στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Γιατί υπάρχει και το θέμα των υποδομών. Χωματερές μονάδες αποτέφρωσης. Τι θα γίνει στο μέλλον με την επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών. we are having. And Εμείς τι κάνουμε που έχουμε μεγάλη δυναμικότητα. Πώς μπορούμε να ε, προχωρήσουμε στην παραγωγή, ε, τη βιολογική παραγωγή ενέργειας κτλ. Θα πρέπει σίγουρα να συνεργαστούμε με τους Δήμους και τις τοπικές κυβερνήσεις και ίσως και κάτι με τις επιδοτήσεις ε, θα πρέπει να γίνει. Thank you very much. And... Ευχαριστούμε πολύ. Απλώς να θυμίσω το χρονοδιάγραμμα 27 Ιουνίου θα ψηφίσει η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια μάλλον τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε κάτι στα διάφορα, απλώς να θυμίσω ότι η επομενη συνεδριαση της Επιτροπής μας είναι 8 Ιουνίου στο Στρασβούργο, καθώς και 16-17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Και τώρα θα σταματήσουμε για λίγα λεπτά για να έρθουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Άγκρη.